Τσεκ had das floor, had the floor for, for zwei Minuten. Δύο λεπτά διακοπή αγαπητοί συνάδελφοι. Okay. Thank you. Thank you, Chair. I will try to get your attention for minutes. Προσπαθήσω για δύο λεπτά να συγκεντρώσω. Να περάσουμε στο επόμενο θέμα. Ευρωπαϊκή Ένωση και Κωσυφοπαίδιο δεν ενθουσιάζει τα πλήθη τόσο πολύ όσο το επόμενο. Αλλά πάση περιπτώσει η Κωσυφοπαίδιο είναι η τελευταία χώρα στα Βαλκάνια που θα έχει μια συμφωνία σταθεροποίησης και σύνδεσης. Είναι το πρώτο βήμα στη διαδικασία ένταξης. Πρόκειται για σφατικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το Κωσυφοπέδιο για πρώτη φορά. Σημαίνει βελτίωση, ενίσχυση του πολιτικού διαλόγου των πολιτικών σχέσεων, σημαίνει επίσης βελτίωση των εμπορικών σχέσεων κλπ. Το Κωσυφοπέδιο θα έχει έτσι περισσότερο πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές για πράγματα όπως είναι το κρασί, που έχει βελτιωθεί τα τελευταία χρόνια μεταξύ άλλων και σημαίνει επίσης και καλύτερες ευρωπαϊκές προδιαγραφές για την προστασία των καταναλωτών, για παράδειγμα κάτι πολύ θετικό για τους πολίτες του κοσμοπεδίου. Επιπλέον θα έχουμε ενισχυμένη συνεργασία, αν μπορώ να χρησιμοποιήσω αυτόν τον όρο, ανάμεσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τη συνέλευση του Κοσμοπεδίου, γιατί δύο φορές το χρόνο θα έχουμε την ε, Επιτροπή Σταθεροποίησης και Σύνδεσης. Όλα αυτά σημαίνουν ότι οι σχέσεις ανάμεσα σε αυτήν την πιο νέα χώρα της Ευρώπης παρόλο που υπάρχουν προβλήματα για στο Σεβούλιο δεν την αναγνωρίζουν όλοι, τα κοινοβούλια και με τη συμφωνία αυτή σταθεροποίηση και σύνδεση μπορούμε να προχωρήσουμε. Είναι θετικά νέα, καλά νέα για τους κατοίκους, τους πολίτες του Κοσμοπεδίου, γιατί είναι ένα σημαντικό βήμα προς την προσχώρησή τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προετοιμάζεται έτσι το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Τώρα, αρχίζουμε στο Κοινοβούλιο. Όσο γίνεται πιο γρήγορα θα ψηφίσουμε στην Ολομέλεια. Αρχές 2016 θα αρχίσει να ισχύει και είμαι πεπισμένη ότι και το επόμενο βήμα που χρειάζονται οι πολίτες του Κοσμοπαιδίου είναι η κατάργηση της υποχρέωσης θεώρησης ε, βίζας. Ελπίζω να γίνει αυτό γρήγορα. Βέβαια το Κωσυφοπέδιο πρέπει να προχωρήσει στην εφαρμογή κάποιων κριτηρίων, αλλά ελπίζω ότι τον επόμενο χρόνο θα είναι αυτό το νέο θετικό για τους πολίτες του Κοσμοπαιδίου στους δύσκολους καιρούς που ζούμε. Έτσι θα τους δώσουμε ελπίδα, θα τους στηρίξουμε και θα τους δείξουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θέλει το κοσυχοπαίδιο να είναι κομμάτι της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτή η Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης, όπως είπα, αποτελεί το πρώτο βήμα με συμβατικές σχέσεις ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το κοσυχοπαίδιο. Καλό σήμα λοιπόν για να προχωρήσουμε. Ελπίζω όλοι να το υποστηρίξουμε, είτε η χώρα σας έχει αναγνωρίσει το κοσμοπέδιο είτε όχι, είναι σημαντικό να πετύχουμε ευρή υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μόνο από την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων. Θα ψηφίσουμε σε λίγες εβδομάδες εδώ, αλλά και αργότερα στην Ολομέλεια. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. ω eh, σκιώδη για το Κωσοφοπέδιο επιτρέψτε μου να παρέμβω κι εγώ. Λοιπόν, εκφράζω την ικανοποίησή μου για τη σύναψη αυτή τη Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση που γίνεται πραγματικότητα σιγά-σιγά. Αποτελεί ένα πολύ σημαντικό στοιχείο για το κοσυφοπαίδιο. Είναι βασικό στοιχείο για την οικονομία της χώρας επίσης όσον αφορά την πρόσβασή της στις αγορές και σε νέες αγορές μάλιστα. Η συμφωνία επιβεβαιώνει ότι το μέλλον του κοσφοπεδίου είναι στην Ευρώπη. Όμως η διαδικασία ένταξης απαιτεί πολιτική βούληση και ηγεσία. Δεν είναι κάτι αυτονόητο. Χρειάζονται μεταρρυθμίσεις από πλευρά της χώρας. Και η κυρία Λούνατσεκ, που είναι συγγήτρια για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, επισκέφτηκε πρόσφατα το κοσυφοπέδιο Και είδαμε Πόση δουλειά έχει κάνει η διοίκηση για να καταπολεμήσει τη διαφθορά που αποτελεί και το κύριο εμπόριο στις δημοκρατικές εξελίξεις. Πρέπει λοιπόν εφαρμοστεί η συμφωνία που μπορεί να μην θέλουν τόσο πολύ όλοι οι ψηφοφόροι, αλλά είναι αποφασιστική σημασία αν θέλουμε οι σχέσεις της χώρας αυτής με τις γείτονες χώρες να ε, γίνουν πραγματικότητα και να είναι κανονικές. Αυτός είναι ο στόχος. Πρέπει όμως να σεβαστούμε και την αντιπολίτευση. Πρέπει να υπάρχει πολιτική βόληση και από τις δύο πλευρές εκατέρωθεν σε αυτή την πορεία. Ευχαριστούμε κύριε Άντακτησον. Οι τρεις που μένουν ένα λεπτό καθένας. Παρακαλώ. Ο κύριος Πατσέρη πρώτα. Ευχαριστώ πρόεδρε. νομίζω ότι μπορούμε να διαπιστώσουμε με τα πρόοδο για την χώρα αυτή και πάνω απ' όλα όσον αφορά το σύμφωνο σταθερότητας και σύνδεσης που υπεγράφει μέσα Οκτωβρίου. Πρόκειται για σημαντικό βήμα όσον αφορά την πορεία της χώρας και του ευρωπαϊκού της μέλλον. και είπαμε ότι έχουμε εξωμάσεις σχέσεων με, το, με την Σερβία ε, αλλά και την λειτουργία δημοκρατία στη χώρα. Υπάρχουν πολλές προκλήσεις που ακόμη απομένει να αντιμετωπιστούν όσον αφορά την ε, οικονομία, τη δημόσια διοίκηση, αλλά επίσης η η υπογραφή αυτής της ε, συμφωνίας με το Κωσικοπαίδιο αφορά την προσχώρηση σε κάποια προγράμματα της Ένωσης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί έτσι πρόκειται να παγιωθούν όλα τα επιδήματα αυτής της χώρας που οδηγούν στην προσέγγιση της προς την Ευρώπη. Ευχαριστώ συνάδελφε Παντσέρη πρόεδρος. Και τώρα το λόγο έχει ο κύριος για ένα λεπτό. Έχετε το λόγο. Είπε η Ρωσία ότι η αναγνώριση του κοσυφοπεδίου σημαίνει ότι ανοίγει το κουτί της Πανδώρας που θα ανοίξει σίγουρα. Ανοίξαν όμως δύο κουτιά Πανδώρας. Έχουμε την εθνοκάθαρση στο κοσυφοπεδίο από τους Σέρβους. Πρόκειται για μια κατάσταση μεταξύ των δύο κοινοτήτων και τώρα αυτό έχει περιοριστεί στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αλλά δυναμηθήσαμε τη συμφωνία του Ελσίνκη για τα σύνορα. Πώς είναι δυνατόν τώρα να λέμε όχι στην υπερδινιστερία, στην ε, υπερδινιστερία, για αυτό την και τι. Και πώς έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Γιατί είπαμε ναι στο κοσικοπέδιο και όχι στην Αμπουχαζία. Ευχαριστώ πολύ αγαπητοί συνάδελφοι. Κύριο Σπίτσουλα, ένα λεπτό παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η Συμφωνία Σταθεροποίηση και Εταιρική Σχέση μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και Κοσμοπεδίου είναι κάνει σαφέ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν αγνοεί την ευρωπαϊκή προοπτική του πιο νέου ευρωπαϊκού κράτου. Αλλά από την άλλη μεριά χρειάζεται η δέσμευση του Κωσυφοπεδίου να κάνει τι απαραίτητε προσπάθειε να ξεπεράσει τα διάφορα προβλήματα που έχει και να προχωρήσει σε βαθιές μεταρρυθμίσεις. Είναι μια ευκαιρία για πολλές ε, ομάδες του πληθυσμού και την κοινωνία του Κωσόβου να προχωρήσει προς την συγχρονικότητα. Βέβαια υπάρχει μεγάλη πίεση προς την κυβέρνηση, αλλά <clears throat> θα πρέπει η διαδικασία αυτή να είναι μια κοινή σύμπραξη όλων των δυνάμεων στη χώρα που έχουν τον ίδιο στόχο η κοινωνία των πολιτών, οι επιχειρηματίες, οι μειονότητες, όλοι πρέπει να κάνουμε την απαραίτητο για να μπορέσει να λειτουργήσει η Συμφωνία Σταθεροποίηση και Σύνδεση. Δεν έχω καμιά αμφιβολία ότι αυτή η συμφωνία θα ευνοήσει και τον διάλογο μεταξύ τη ε, Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Πριστίνα, αλλά και μεταξύ τη Πριστίνα και του Βελιγραδίου. Η περιφερειακή συνεργασία στα Δυτικά Βαλκάνια λοιπόν θα μπορέσει να ευνοηθεί και να ξεπεραστούν τα προβλήματα ασφαλεία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέει και ο πρόεδρο Μπροκ. <clears throat> Θέλω να σας αναφέρω ότι η προθεσμία κατάθεση τροπολογιών 20 Νοεμβρίου θα γίνει συζήτηση στις 19 Νοεμβρίου και μετά στην 2η Δεκεμβρίου θα συνεχίσουμε και στις 14 Δεκεμβρίου πρέπει να, πάρουμε, να κάνουμε την ψυχοφορία στην Επιτροπή μας. Ελπίζω να συμφωνείτε με αυτό το χρονοδιάγραμμα <clears throat> για να μπορέσουμε να φέρουμε το θέμα αυτό στην Ολομέλεια. Έχουμε τώρα στο επόμενο σημείο τη διάταξη που είναι η ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, τον κύριο Φρανκ Βάλτερ Στάινμαερ, ο οποίος έρχεται κατευθείαν από το Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών και μπορεί να μας πει για τα θέματα της αντιμετώπισης της τρομοκρατίας μετά από το, τις επιθέσεις στο Παρίσι. Θα, μας, θα αναφερθεί όμως επίσης και στα θέματα της Συρίας και της ε, Ουκρανίας και επίσης η Γερμανία αναλαμβάνει την προεδρία του, ΟΑ, του ΟΑΣΕ, οπότε και αυτό είναι ένα περαιτέρω θέμα το οποίο έχει μεγάλο ενδιαφέρον και σας δίνω μέσα στο λόγο κύριε Στάνιμαρ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θέλω και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση που μου απευθύνατε. <clears throat> Με μεγάλη χαρά έρχομαι ενώπιον σας γιατί νομίζω ότι είναι απαραίτητο ο διάλογος και οι επαφές μεταξύ ε, εμού και της Επιτροπής σας. Θέλω να σας ευχαριστήσω επίσης και για την ε, υποστήριξη που έχουμε λάβει από την Επιτροπή σας για σημαντικά θέματα όπως είναι η ανατολική εταιρική σχέση τους τελευταίους μήνες και δεν θα λησμονήσω να αναφερθώ τις προσπάθειες που έχουν καταβάλει τα μέλη της Επιτροπής σας για να ξεπεραστεί το η κατάσταση αδιεξόδου η οποία είχε δημιουργηθεί στην Αλβανία και που δεν θα μπορούσε να ξεπεραστεί χωρίς τις προσπάθειες που έχετε καταβάλει για να δημιουργηθεί ένα κλίμα περισσότερης εμπιστοσύνης. Θέλω λοιπόν να σας ευχαριστήσω και για την ευκαιρία να παρουσιαστώ ενώπιόν σας και αυτό φυσικά σε μια χρονική στιγμή που είναι ιδιαίτερα ιδιαίτερη που έχει σημαδευτεί από, τις, ε, από τα τραγικό, τραγικά γεγονότα του Σαββατοκύριακου στο Παρίσι. Εκείνη τη μέρα εγώ ο ίδιος ήμουνα παρόν στο Παρίσι, ήμουνα στο Stade de France, στο ίδιο το γήπεδο και ο στόχος ήταν να παρίσταμε στον αγώνα των ε, φιλικών των εθνικών ομάδων των δύο χωρών, της Γερμανίας και της Γαλλίας. Και ενώ θα έπρεπε να είναι ένα ορταστικό γεγονός, αντιμετωπίσαμε μια πραγματική τραγωδία. Δεν ήτανε κάτι σαν την κατάρριψη ή σαν την πτώση ενός ε, αεροσκάφους. Όπως η περίπτωση του German Wings όπου υπήρξε μια πολύ μεγάλη ε, συμμετοχή και των δύο πλευρών για να μπορέσουν να αντιμετωπιστούν τα θύματα. Σε αυτή την περίπτωση είχαμε μια πραγματικά ανοιχτή τρομοκρατική επίθεση που εκδηλώθηκε σε διάφορα σημεία των Παρισίων. Και εμείς κρατήσαμε ενός λεπτού σιγή στο Συμβούλιο των Υπουργών εις μνήμη των θυμάτων. Αλλά τώρα η κατάσταση μετά από τις τρομοκρατικές επιθέσεις έχει δημιουργήσει και άλλα ερωτήματα. Θα πρέπει να αντλήσουμε τα συμπεράσματα από αυτή την κατάσταση. Αυτό που είναι απαραίτητο είναι να μπορέσουμε να θέσουμε τα σωστά ερωτήματα και είναι πολύ σημαντικό να δούμε και πόσες στρατιωτικές δυνάμεις θα μπορέσουν να διατεθούν από τα κράτη-μέλη για να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες προστασίας. Δεν μπορώ τώρα να σας δώσω πραγματικές λεπτομέρειες για όλα αυτά τα θέματα, αλλά είναι σαφές πώς θα πρέπει να δράσουμε για να αντιμετωπίσουμε την τρομοκρατία. Δεν είναι εύκολες οι απαντήσεις. Μετά από το Παρίσι τα πράγματα είναι ακόμα πιο δύσκολα. Εμείς ως ε, Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση της Γερμανίας θα συνεχίσουμε να είμαστε απόλυτα προσιλωμένοι στην προσπάθεια αντιμετώπισης της τρομοκρατίας. Είναι πολλές οι χώρες οι οποίες έχουν διαδηλώσει την θέλησή τους να συμμετάσχουν σε αεροπορικές επιδρομές κατά της, ε, του Ισλαμικού κράτους από την πλευρά της Γερμανίας. Εμείς έχουμε συμβάλει σημαντικά στο να εκπαιδεύσουμε αυτούς οι οποίοι αγωνίζονται στο έδαφος τους Πεσμεργά από το Βόρειο Ιράκ, οι οποίοι μάχονται κατά του Ισλαμικού κράτους. Η Γερμανία έχει παίξει σημαντικό ρόλο για να τους εκπαιδεύσουμε και παρά τις ε, συζητήσεις οι, οποία, οι οποίες έλαβαν χώρα στη γερμανική κοινή γνώμη έχουμε αποφασίσει να δώσουμε εκπαίδευση και εξοπλισμό στους Πεσμεργά όχι μονάχα για να μπορέσουν να κρατήσουν την γραμμή του μετόπου αλλά για να μπορέσουν να δράσουν αποτελεσματικά κατά του Ισλαμικού κράτους και ελπίζω ότι αυτή η διαδικασία θα συνεχιστεί τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Εμείς θα συνεχίσουμε φυσικά την υποστήριξή μας προς αυτούς και είμαστε σε στενή επαφή με τους υπεύθυνου των στρατιωτικών αυτών δυνάμεων, των Πεσμεργά και έχουμε τακτικές αναφορές για αυτούς σε σχέση με τις ανάγκες που πρέπει να αντιμετωπιστούν και στις οποίες πρέπει να συμβάλλουμε. Αυτό σα το λέω γιατί πιστεύω ότι είναι κάτι το οποίο γνωρίζετε ότι πρέπει να συνεχιστεί ο αγώνα κατά του Ισλαμικού κράτους σε στρατιωτικό επίπεδο, αλλά φυσικά γνωρίζουμε όλοι ότι δεν μπορούμε μόνο με στρατιωτικά μέσα να αντιμετωπίσουμε οριστικά το πρόβλημα της τρομοκρατία. Οπότε αυτό με φέρνει στο δεύτερο σημείο το οποίο έτυχε συζήτηση κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου των Υπουργών Εξωτερικών. Ήταν το θέμα του, της Συρίας. Πώς μπορούμε να μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε την ε, επίλυση σε πολιτικό επίπεδο της ε, σύραξης στην Συρία. Όποιος γνωρίζει τη Μέση Ανατολή και εσείς ιδιαίτερα το ξέρετε, όποιος ε, λαμβάνει το λόγο και κάνει μια δήλωση για τα θέματα αυτά, θα πρέπει να είναι πολύ προσεκτικός να μην δημιουργήσει ένα φρούδο κλίμα εφορίας και αισιοδοξία. Οι συζητήσεις οι οποίες έγιναν προηγουμένως στη Βιέννη για το θέμα της Συρίας έφεραν κάποια αποτελέσματα τα οποία ήταν λιγάκι απρόσμενα. απρόσμενα πρώτα απ' όλα γιατί καταρχήν έγινε για πρώτη φορά δυνατό όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να είναι παρόντα. Το να πούμε ότι θα ήταν δυνατόν πριν από τρει μήνε να συζητήσει η Ρωσία μαζί με τις ΗΠΑ για τη Συρία και να βρεθούν στο ίδιο τραπέζι, αυτό θα θεωρούσαμε ότι ήταν απόλυτα αδύνατο. Επίσης, κανείς δεν θα μπορούσε να πιστέψει ότι θα μπορούσε το Ιράν και η Σαουδική Αραβία να βρίσκονται στο ίδιο τραπέζι και να διαπραγματεύονται για το ίδιο αυτό θέμα. Το γεγονός ότι αυτό επετεύχθη είναι μια τεράστια επιτυχία, μια τεράστια πρόοδος που έχει αφεαυτής μεγάλη αξία. Αυτό το οποίο πρέπει να προσπαθήσουμε τώρα να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ένα μόνιμο σχήμα διαπραγμάτευσης σε επίπεδο στρογγυλής τράπεζας με όλους τους εμπλεκόμενους σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό λοιπόν μπορούμε να προχωρήσουμε και πέραν της ε, συμφωνίας που οδήγησε στη δήλωση πριν από δύο εβδομάδες ότι δεν θέλουμε να υπάρξει, δεν μπορούμε να δεχτούμε τον κατακαιρματισμό της Συρίας, ότι θα διατηρηθεί η εδαφική ακαιρεότητα της Συρίας και ότι στο μέλλον η Συρία θα πρέπει να έχει μια τέτοια μορφή ώστε να εξασφαλίζει την συμβίωση όλων των εθνοτικών και θρησκευτικών ομάδων και όχι την αντιπαράθεσή τους. Για ορισμένους αυτό φαίνεται ότι είναι μια ουτοπία. Αλλά ε, με τη συμμετοχή του Ιράν και με τη συμμετοχή της Ρωσίας κατέστη δυνατόν πέραν των αρχών που διαδηλώσαμε να χαράξουμε και ένα οδικό χάρτη να συμφωνήσουμε για μια διαδικασία η οποία θα οδηγήσει πρώτα σε μια ανακοχή και δεύτερον τη δημιουργία μιας μεταβατικής κυβέρνησης στη Συρία και τρίτον την ε, διατύπωση ενός συντάγματος στη Συρία που θα οδηγήσει σε εκλογές στη Συρία. Αυτούς τους τέσσερις στόχους λοιπόν μπορούμε να επιτύχουμε με, σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα χάρη στην ε, συμφωνία που επετέφθη στη Βιέννη. Πρώτα απ' όλα φυσικά πρέπει να προετοιμάσουμε μια ανακοχή και θα γίνουν και πάλι συζητήσεις όπου θα συμμετέχουν εκπρόσωποι της κυβέρνησης αλλά και της αντιπολίτευσης με στόχο σε αυτές τις διαπραγματεύσεις να μπορέσει να εξασφαλιστεί μια ανακοχή. Επομένως ο στρατός της Συρίας και οι ένοπλες δυνάμεις της αντιπολίτευσης θα πρέπει να σταματήσουν να βρίσκονται σε ένοπλη αντιπαράθεση. Δεύτερον, μέσα σε έξι μήνες από σήμερα θα πρέπει να δημιουργηθεί μια μεταβατική κυβέρνηση και τρίτον η διαδικασία αυτή πρέπει να δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε μέσα σε 18 μήνες από σήμερα να γίνουν εκλογές. Το ερώτημα του τι θα γίνει με τον Μπασάρ Αλασάντ, αυτό είναι ένα θέμα το οποίο παραμένει ακόμα ασαφές στο κοινό έγγραφο. Είναι φανερό ότι βρίσκονται στην τράπεζα των διαπραγματεύσεων και οι υπέρμαχοι του Ασάντ και αυτοί οι οποίοι θεωρούν το μέλλον της Συρίας οπωσδήποτε δεν μπορεί να περιλαμβάνει τον Ασάντ. Δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να καταλήξουμε σε ένα οριστικό αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο είναι σημαντικό τώρα η, η πολιτική διαδικασία να κινήσει <clears throat> και να μπορούμε το ταχύτερο δυνατόν να έχουμε τις προϋποθέσεις για μια ανακοχή. Όπως βλέπουμε εμείς από την ευρωπαϊκή πλευρά, είναι πολύ σημαντικό όχι μονάχα η Ευρώπη και η Ευρωπαϊκή Ένωση να συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία, είναι επίσης και η δική μας θέληση και επιθυμία αυτή η διαδικασία να τεθεί υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε δεχτεί και το έχουμε συμφωνήσει το προηγούμενο Σάββατο. Εάν μπορέσει να υπάρξει λοιπόν αποκλιμάκωση στην Συρία, θα έχει ανοίξει ή τουλάχιστον θα είναι ορατός ο δρόμος για μια πολιτική λύση και επομένως θα μειωθεί και η ανάγκη για αντιπαράθεση με το Ισλαμικό κράτος και επομένως θα αυξηθεί και η ευρωπαϊκή ασφάλεια. Έρχομαι τώρα σε ένα άλλο θέμα που συζητήθηκε, το θέμα της Ουκρανίας. Και εδώ δεν υπάρχει λόγος να πανηγυρίσουμε. Συνεχίζονται και εκεί οι προσπάθειες για να αντιμετωπιστεί η αντιπαράθεση εκεί και δεν πρόκειται εγώ να ωρεοποιήσω την κατάσταση στην Ουκρανία. Πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται από την εφαρμογή της συμφωνίας του Μίνσκ. Έχουμε ακόμα παραβιάσεις της κατάπαυσης του πυρός που έχουν λάβει χώρα και τις τελευταίες μέρες έχουν αυξηθεί. Από το, την 1η Σεπτεμβρίου όμως σε μεγάλο βαθμό μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι λειτουργεί αυτή η διαδικασία, είναι απαραίτητο να συνεχίσουμε την ε, προσπάθειά μας να εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει πλήρης τήρηση της κατάπαυσης του πυρός. Υπάρχει μια διαδικασία απόσυρσης των ελαφρών όπλων και σε μια συνάντηση στο Βερολίνο έχουμε αποφασίσει ότι μετά από την απόσυρση των ελαφρών όπλων θα ακολουθήσει και η απόσυρση των βαρέων όπλων. Πρέπει να προχωρήσουμε στη συνέχεια σε αποναρκοθέτηση. και επομένως να μπορούν οι άνθρωποι να διακινούνται ελεύθερα στην Ουκρανία χωρίς να φοβούνται ότι μπαίνουν σε ναρκοπαίδια ή σε γραμμές ένοπλης αντιπαράθεση. Επίσης μας έχει απασχολήσει το θέμα της ανθρωπιστικής ανάγκης βοήθειας. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή πολύ περιορισμένος αριθμός οργανώσεων που λειτουργούν στην ε, Ουκρανία πέραν του Ερυθρού Σταυρού Επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρχει και η ανταλλαγή των εχμαλώτων, κάτι το οποίο έχει αποφασιστεί ήδη. Είναι πολύ μικρό ο αριθμό ο οποίος έχει ανταλλαγή μέχρι τώρα, αλλά υπάρχουν χιλιάδες ακόμα που βρίσκονται στις αντίστοιχε ε, φυλακές και κέντρα κράτηση. Έχουμε πετύχει λοιπόν αυτές τις περιορισμένες επιτυχίες για τη Ρωσία. Η Ρωσία είναι αυτή η οποία προκάλεσε αυτήν την κρίση και για πολύ καιρό έκανε ό,τι μπορούσε ώστε οι διαπραγματεύσεις στο Παρίσι και στο Βερολίνο να μην προχωρήσουν ρούπι. Είναι απαραίτητο λοιπόν να τονίσω ότι υπήρξε κάποια μετακίνηση του ενδιαφέροντος στη Ρωσία προς την Συρία και η Ρωσία για αυτό το λόγο έχει λιγότερη έμφαση στην ε, σύγκρουση της ε, Ουκρανίας. Δεν έχει σημασία ποιοι είναι οι λόγοι οι οποίοι έχουν οδηγήσει σε κάτι τέτοιο. <clears throat> Αλλά η Ρωσία τον τελευταίο καιρό έχει δείξει μια πιο ε, επικοδομητική ε, στάση. Ευτυχώς και οι αυτονομιστές έχουν αναβάλει τις εκλογές οι οποίες θα λάμβαναν χώρα στο ανατολικό τμήμα της Ουκρανίας και έτσι έχει αποφευθεί να παρακαμφθεί τελείως η συμφωνία του Μίνσκ. Μπορούμε, πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να υποστηρίξουμε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι καθόλου αυτονόητη, δεν μπορεί να προχωρήσει μόνη της. Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε μια συμφωνία και τον επόμενο Μάρτιο που θα γίνει συνάντηση στην Ορμανδία. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει να αντιμετωπίσει και το θέμα της ε, συνέχισης ή μη των κυρώσεων. Δεν έχει ξεκινήσει καθόλου η συζήτηση ακόμα μέχρι στιγμή. Όλα αυτά όμως εξαρτώνται από το βαθμό εφαρμογής της διαδικασίας του Μίνσκ. Θα πρέπει λοιπόν να συνδέσουμε τις ε, κυρώσεις και την διατήρηση ημί με την επιτυχία της εφαρμογής του, της συμφωνίας του Μίνσκ η οποία θα πρέπει να οδηγήσει σε εκλογές και την ε, επαναφορά του ελέγχου των συνόρων στις Ουκρανικές αρχές. Και κάτι τελευταίο και πάρα πολύ σύντομο, ξέρετε ότι σε ό,τι αφορά <clears throat> την παρακολούθηση και επαλήθευση την ε, αποστολή επαλήτευσης η ΟΣΑ, η ΟΑΣΕ, συγγνώμη, έχει παίξει σημαντικό ρόλο. Η Ελβετική Προεδρία έχει παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο για να μπορέσει να γίνει δυνατό να χρησιμοποιηθεί ε, η οργάνωση αυτή, ο ΑΣΕ, Εμείς τώρα μετά από τη Σερβία τον επόμενο χρόνο, από τον Ιανουάριο, θα αναλάβουμε την προεδρία της ΟΑΣΕ, γνωρίζοντας πάντα ότι είναι μια δύσκολη κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΟΑΣΕ, ότι η οι αντιπαραθέσεις και οι συγκρούσεις στην Ουκρανία αντανακλώνται και στο εσωτερικό της ε, ΟΑΣΕ, αλλά Πρέπει να τονίσω ότι αυτός ο οργανισμός είναι ένας από τους λίγους φορείς οι οποίοι έχουν έχουν επιβιώσει κατά κάποιο τρόπο του τέλους του ψυχρού πολέμου και έχουν παίξει σημαντικό ρόλο και μετά από τις κρίσεις της Μολδαβίας και της Γεωργίας είναι από τους λίγους φορείς λοιπόν που είναι λειτουργικός και μπορεί να έχει ένα πραγματικό αντίκτυπο. Γι' αυτό αποφασίσαμε και εμείς παρά τις ε, ανησυχίες και τις αντιρρήσεις που ε, είχαν εκφραστεί να αναλάβουμε την Προεδρία του ΟΑΣΕ. Έχουν προχωρήσει, προχωρήσει οι προετοιμασίες και θα είναι σίγουρο ότι δεν θα περιοριστούμε μονάχα στα θέματα της ε, διαμεσολάβησης στην Ουκρανία, αλλά θα αντιμετωπίσουμε και τα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του αντισημιτισμού με τον πρέποντα τρόπο. Αυτά είναι λοιπόν οι αρχικές μου παρατήρησεις και είμαι έτοιμος να προχωρήσω στη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ και ο Πρόεδρος. Εγώ έχω να θέσω προσωπικά ένα ερώτημα. Θέλω τώρα να ζητήσω πρώτα να περιοριστούν οι συντονιστές σε ένα λεπτό και οι υπόλοιποι ομιλητές σε ένα λεπτό. Ζητώ την κατανόησή σας για να μπορούμε να έχουμε την ευκαιρία όλοι να εκφράσουμε τα, τις απόψεις μας. Το δικό μου θέμα, το δικό μου ερώτημα είναι, είπατε ότι έχετε ένα χρονοδιάγραμμα για τη Συρία, μια διαδικασία 6 μηνών και μια διαδικασία 18 ετών μέχρι τις εκλογές. Υπάρχει λοιπόν η δυνατότητα, εάν ευδοκιμήσει αυτή η διαδικασία, να έχουμε μια γενική συμμαχία κατά του Ισλαμικού κράτους. Αυτό είναι το ερώτημά μου. κύριος Φρέντα τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε κύριος Φρέντα. Κύριε Υπουργέ, σας περιμέναμε για να συζητήσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η εξωτερική μας πολιτική. Στο μεταξύ βέβαια οι επιθέσεις κατά του Παρισιού την Παρασκευή που μας πέρασε έδωσαν βέβαια άλλη απόχρωση στη συνάντησή μας αυτή. Φυσικά και είμαστε αλληλέγγυοι με τους Γάλλους φίλους μας και με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες που έχασαν δικούς τους στις επιθέσεις αυτής Βέλγοι, Βρετανοί, Ισπανοί, Ιταλοί, Ρουμάνοι που όλοι αυτοί ήταν θύματα αυτών των φρικτών επιθέσεων. Η αλληλεγγύη όμως πιστεύω ότι πρέπει να πάει πέρα από τις δηλώσεις. Νομίζω ότι στη συνθήκη της Λισαβόνας υπάρχει μια ρήτρα αλληλεγγύης, είναι το άρθρο 222, το οποίο τι λέει, λέει ότι εάν αποτελεί αντικείμενα τρομοκρατικής επίθεσης μια χώρα μέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση, τότε χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που έχει στη διάθεσή της, ακόμη και στρατιωτικά, για να προστατεύσει τους δημοκρατικούς θεσμούς και, για να βοηθήσει την λόγω χώρα μέλος στο δαφός της. Ποια είναι η αποψή σας λοιπόν για τη χρησιμότητα αυτή, να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή σε αυτή την περίπτωση το άρθρο 222, το οποίο αναφέρεται σε ρήτρα αλληλεγγύης. Και μία ερώτηση για την ε, αντιπαράθεση στην Ουκρανία και την άρση των κυρώσεων. Ποια είναι η γνώμη σας για την άρση κυρώσεων πριν να φύγει από την Κρυμαία η Ρωσία. Πιστεύετε ότι είναι λογικό να αρθούν οι κυρώσεις πριν να φύγει από την Κρυμαία η Ρωσία. Μπορούμε να εξηγήσουμε κάτι τέτοιο στους πολίτες μας και πώς. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Υπουργέ, Μάιερ, εκ μέρους της πολιτικής μου ομάδας, θέλω να σας ευχαριστήσω πρώτα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Επίσης, θέλω να σας ευχαριστήσω και αυτά τα οποία έκανε η κυρία Μογκερίνη, η ύπατη εκπρόσωπο μας. Μετά από τις πρώτες επιτυχίες που οδήγησαν στη συμφωνία με το Ιράν, έχει συνεχίσει με τρόπο συνεπή και συνεκτικό <clears throat> τις προσπάθειες της σε διπλωματικό επίπεδο και φυσικά είναι απαραίτητο να μπορέσουμε να βρούμε μια λύση για τα θέματα της Συρίας. Θέλω επίσης να σας ευχαριστήσω όπως και την κυρία Μογκερίνη για τις συζητήσεις που διοργανώσετε στο Παρίσι και στο Βερολίνο. Ξέρουμε ότι το γεγονός ότι η Ρωσία έχει κρατήσει μια πιο επικοδομητική στάση. Αυτό είναι φυσικά μια αρχή, δεν είναι επαρκές από μόνο του, αλλά έτσι λειτουργεί και η δημοκρατία με μικρά βήματα, κάτι το οποίο ορισμένοι άλλοι δεν έχουν κάνει ακόμα. Και δεν θα αναφερθώ φυσικά καθόλου σε στρατιωτικές λύσεις για τα προβλήματα αυτά οι κυρώσεις που έχουν επιβληθεί κατά της Ρωσίας και κατά την άποψη της δικής μου πολιτικής ομάδος μπορούν να αρθούν μονάχα όταν υπάρξουν σημαντικές πρόοδοι στην εφαρμογή της διαδικασίας του Μίνσκ. Δεν έχουμε επιλέξει με αφαίρετο τρόπο αυτές τις κυρώσεις, επομένως δεν μπορούμε αφαίρετα να τις άρουμε. Θα πρέπει να υπάρχουν συγκεκριμένες προϋποθέσεις. Όσο πιο οργανωμένη και προβλεπτή είναι αυτή η διαδικασία, τόσο καλύτερα και για όλους. Ναι. Και μια μονάχα τελευταία φράση. Ανεξάρτητα από την άρση των κυρώσεων, τη μείωση των κυρώσεων, θα ήθελα να ρωτήσω κατά πόσο θα μπορούσε να αφαιρεθεί ο, η μαύρη λίστα, να αφαιρεθούν μάλλον από τη μαύρη λίστα που έχει διατυπωθεί. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχουμε το άρθρο 42, παράγραφο 7, όσον αφορά την τελική βοήθεια σε περιπτώσει επιθέσεις που ούτε ε, αυτό συζητήθηκε να εφαρμοστεί. Και έχουμε και το άρθρο 5 του ΝΑΤΟ. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα χρησιμοποιηθούν οι δυνατότητε που Τώρα για το Σέγγεν, ξέρω ότι δεν είναι αρμοδιότητά σα, αλλά ε, για, για πέστε μου, κάποιοι από τους τρομοκράτες του Παρισίου ε, εμφανίστηκαν ως πρόσφυγες από τη Συρία και λένε ότι έφεραν ε, όπλα από τις Βρυξέλλες μια που δεν υπάρχουν πραγματικά σύνορα ε, γαλλοβελγικά και τι λέτε, τι θα γίνει ε, γιατί ο καγκελάριο της Γερμανίας έχει πει ότι θα πρέπει να δώσει με ανοιχτά σύνορα πλήρες άσυλο σε τους ε, Σύρους. Επίσης η κυβέρνηση της Βαβαρίας απειλεί να ξαναρχίσει τους συνορικούς ελέγχους, κάτι το οποίο έχει την αρμοδία να το κάνει. Και επίσης τι γίνεται όσον αφορά τις ε, ελληνικές αρχές που κάποιον συνέλαβαν από το Μαυροβούνιο και ε, αυτός ενώ είχε πριν περάσει από την Αυστρία τον άφησαν ελεύθερο και άρα έχουμε κακή, ε, κακή συνεννόηση. Μπορούμε να αποσυνδέσουμε την Ρωσία από τις ε, κυρώσεις για την Ουκρανία για το θέμα της Συρίας, για αυτό που κάνει τώρα η Συρία, να της δώσουμε δηλαδή κάποιο είδους αμνηστία εάν συμφωνεί η Τεχεράνη και η Τουρκία ας πούμε για τους Πεσμεργά τώρα Είχαμε έρθει σε επαφή πρόσφατα και λέγανε ότι έχουν κάποιες επιφυλάξεις για ποσότητα και ποιότητα των όπλων. Εσείς είπατε ότι έχουν κάτι αντιαρματικά, έχουν τα δικά τους όπλα, αλλά τι μπορούμε να κάνουμε τόσο σε αυτούς τους γενναίους μαχητές που εκεί μάχονται ε, το Ισλαμικό κράτος να τους δώσουμε αυτά τα οποία χρειάζονται. Καλώ ήρθατε κύριε Υπουργέ. Θα ήθελα εξ ονόματος της ε, ομάδος του Άλντε να αναφερθώ και στο θέμα του Σέγγεν από μια διαφορετική οπτική γωνία. Για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την κρίση των προσφύγων και αυτό φυσικά δεν αφορά ε, την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας και του εγκλήματος, είναι απαραίτητο να έχουμε έλεγχο των εξωτερικών συνόρων του Σέγγεν, όχι να τα κλείσουμε αλλά να τα ελέγξουμε τι πρωτοβουλίες θα αναλάβει η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση Γερμανίας ώστε να εφαρμόσει σωστά τον έλεγχο των συνόρων. Αυτό είναι το πρώτο μου ερώτημα. Δεύτερο, για την ε, Συμφωνία του Μίνσκ. Η ε, εποπτεία των συνόρων της Ουκρανίας με τη Ρωσία είναι απαραίτητη. Χωρίς τον έλεγχο των συνόρων της από την πλευρά της ε, Ουκρανίας πιστεύω ότι δεν πρέπει να υπάρξει άρση των κυρώσεων. Συμφωνείτε με αυτή την άποψη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κυρία η κυρία Λέζιν που ήρθατε για να απαντήσετε τα ερωτήματά μας εξ ονόματος της ε, ομάδας της Ευρωπαϊκής Ενωτικής Αριστεράς. Θέλω να σας θέσω και ένα ερώτημα για το Αφγανιστάν. Η Γερμανία έχει ήδη μια εκστρατεία που έχει οργανώσει στο Αφγανιστάν με αφήσει, με ενημερωτικέ ε, ε αφήσει και πλακάτ για να προειδοποιήσει τους πολίτες να μην θέτουν τους εαυτούς τους στα χέρια των διακινητών και να κινούνται προς την Ευρώπη. Ο κύριος Μπάικη είπε ότι οι γερμανικές αρχές ζητήσα, από τις γερμανικές αρχές να δεχτούν πρόσφυγες από το Αφγανιστάν και να μην τους αποθήσουν για λόγους ασφάλειας. Ποια είναι η δική σας θέση για την απότηση προσφύγων από το Αφγανιστάν στην Γερμανία. Και επίσης πώς θα εξασφαλιστεί ότι η αποστολή του ΝΑΤΟ θα μπορούσε να έχει μια πραγματική εντολή ε, μετά από τη δράση των, του γερμανικού στρατού στο Αφγανιστάν. Και πιστεύετε ότι θα πρέπει να συνεχιστεί η δράση του ΝΑΤΟ στο Αφγανιστάν ή όχι. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ τον κύριο Στάινμαερ για την έλευσή του στην Επιτροπή μας για τα θέματα της Συρίας και μιλώ εξ των Πρασίνων. Ξέρουμε φυσικά ότι θα πρέπει να υπάρξει αυτό το, αυτός ο οδικός χάρτης για τη Συρία που πρέπει να εφαρμοστεί. Είπατε στην αρχή ότι δεν μπορείτε να ξέρετε μέχρι πού θα μπορέσει να αντιμετωπιστεί αυτό το σύνολο θεμάτων, αλλά είναι γεγονός ότι έχουμε να αντιμετωπίσουμε μια σειρά από εγκλήματα κατά της ανθρωπότητος πιστεύετε ότι έστω σε ένα μεσοπρόθεσμο επίπεδο θα μπορέσουν να έρθουν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι για αυτά τα εγκλήματα. Μετά από τη συνάντηση της Βιέννης είπατε ότι μεταξύ της ε, Ρωσίας και των κρατών του Περσικού κόλπου υπήρξε μια έλλειψη συμφωνίας για το ποιες ομάδες, ένοπλες ομάδες θα πρέπει να θεωρηθούν ως τρομοκρατικές. Υπάρχει κάποια προσπάθεια να γεφυρωθούν αυτές οι θέσεις και ακριβώς για ποιες ομάδες συζητήθηκε το θέμα αυτό. Και επίσης λαμβάνεται η δυνατότητα η Διεθνής Ομάδα Υποστήριξης της ε, Συρίας να αντιμετωπίσει τις ανάγκες του πληθυσμού σε περιοχές οι οποίες ελέγχονται από το Ισλαμικό κράτος. Ευχαριστώ. Έχει κλείσει ο κατάλογος των αγορητών. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Πες μας τι γίνεται με την ελεύθερη διακίνηση. Πιστεύετε ότι σχετικά με αυτό θα πρέπει και τα κράτη-μέλη να μπορούν να λάβουν κάποιες ε, αποφάσεις εάν υπάρχει διακύβευση των συγχρόνων τους. Γιατί είδατε είχαμε αυτά τα τρομερά γεγονότα στο Παρίσι. Οπότε τώρα ε, θέλει να κλείσει τα σύνορα η γαλλική κυβέρνηση και άλλες κυβερνήσεις να ξαναρχίσουν τη συνεργούς ελληνικούς. Άρα έχουμε το τέλος του Σέγγεν. Και τι έγινε με εκείνον τον ε, Μαυροβούνιο. Του βρήκατε 8α47, χειροβομβίδες, εκρηκτικά, τέλος πάντων πυρομαχικά και τι γίνεται. Αυτό δεν ήταν ματίωση κάποιας ε, τρομοκρατικής ενέργειας. και ένα δορυφόρο, είδε από το κινητό του ότι θα πήγαινε στο Παρίσι αυτό που το οδηγούσε. Λοιπόν, τι γίνεται με το Σέγγεν και σχετικά με αυτό. Είπε η κυρία Μέρκελ, ότι πρέπει να υπάρχει ενωσιακό στρατό και ο Κάμερον θα πρέπει να το δεχθεί ε, πέραν αυτών των ε, ονομαστικών ε, μεταρρυθμίσεων και έτσι να παραμείνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την συνήκη της Λισαβόνας. Δεν θα πρέπει κάποια στιγμή να την αναθεωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τι γίνεται επίσης όσον αφορά την χρηματοδότηση αυτού του ε, ενωσιακού στρατού. Αν δεν είναι ο λαός γιατί θα πρέπει να κατευθύνουν τα στρατικά και πάλι οι Γερμανοί. Και τελικά εσείς δεν μπορέσατε στην Λιβύη το 2011 να κάνετε κάτι στο Ιράκ για να υποστήσετε κάτι τις προσπάθειες που έγιναν εκεί. Ντονζό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Υπουργέ. Είμαι ο πρώτος Γάλλος που λαμβάνω το λόγο σήμερα σε αυτή τη συνεδρίαση και γι' αυτό και σας ευχαριστώ για τα λόγια ελληνικής αλλά και όλους τους συναδέλφους της ε, ομάδας που και το Σαββατοκύριακο αλλά και σήμερα εξέφρασαν την υποστήριξη προς το γαλλικό λαό που τόσο σκληρά χτυπήθηκε, ήταν τόσο τραυματικά αυτά που γίνανε την Παρασκευή το βράδυ στο Παρίσι, το Παρίσι χτυπήθηκε, αλλά δεν είναι η πρώτη ε, ε πόλη στην Ευρώπη που το παθαίνει αυτό. Έχουν ήδη χτυπηθεί το Μαδρίτη, το Λονδίνο, αλλά δεν θα είναι ούτε η τελευταία δυστυχώ και λόγω ακριβώ του μεγέθου αυτή τη απειλή. Είπατε κύριε ε, Υπουργέ ότι δεν μπορεί να υπάρχει αντίδραση παρά μόνο στρατιωτική αντίδραση. Τι να σας πω, αλλά από την άλλη μεριά έχουμε αυτές τις αιστείες αστάθειες είναι πάρα πολλές. Ποτέ δεν ήταν τόσες πολλές κοντά στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αφρική και στο κέρας της Αφρικής και στην Κεντρική Αφρική και βεβαίως και στην εγγύση Ανατολή αλλά και προς Ανατολάς της Ευρώπης. Οπότε λένε οι συμπατριώτες μου ότι πολλές φορές η Γαλλία ε, είναι μόνη ε, και βρίσκεται στις πρώτες γραμμές αυτής της ε, μάχης. Αλλά η Γερμανία είναι πρωταθλήτρια τώρα στην Ευρώπη και άκουσα στο μόναχο την ομιλία σας, ήταν ε, ε, ε πολύ θαραλευτά που είπατε με τον Γκάου και τον Ντελάγεν και είπατε ότι θα πρέπει να λάβει η Γερμανία πιο δυναμικό ρόλο στη διεθνή σκηνή. Όμως σήμερα τι θα κάνετε οι, οι Γάλλοι θα θέλανε η πιο μεγάλη ευρωπαϊκή χώρα να δείξει ακόμα πιο πρακτικά, ακόμα πιο ενεργά την ελληνική της στη διεθνή σκηνή. Πρόεδρος. Ένα λεπτό, αλλά πρώτα πρώτα, ένα λεπτό έχει ο καθένα είπαμε. Αλλά πρώτα ο κύριο Παντσέρη, σα ευχαριστώ με που ήρθατε κύριε Υπουργέ. Έχω δύο ερωτήσει να σα υποβάλω. Πρώτα πρώτα, ε, γιατί αντιλήφθηνα ότι στην ε, συζήτηση ε, ε Όντω έχουμε συνειδητοποιήσει όλοι το ότι είσαστε στην ηγεσία του γραμμή τη Ευρώπη και όσον αφορά ε, την εξωτερική μας πολιτική, για την ε, πρόκληση που έχουμε έτσι ε, πρέπει να κάνουμε, την πρόκληση της τρομοκρατίας. Έχουμε τώρα και κάποιους διεθνείς παρατηρητές στη συνάντηση της Βιέννας και είπαμε ότι θα πρέπει κάτι να γίνει κατόπιν των κινήσεων της Ρωσίας στην Συρία. Καλό, για πέστε μας, άπαξ και είπαμε ότι οι στόχοι για την Συρία είναι το κράτο κράτος θα πρέπει μετά να έχουμε κάποια μεταβατική κατάσταση για να αντικαταστεί τον Άσαντ εσείς τι θεωρείτε θα πρέπει να γίνει, θα πρέπει να είναι πρώτος στόχος ε, το Ισλαμικό κράτος. Ευχαριστώ. Κύριε κύριε Υπουργέ, σας βεβαιώνω ότι όλοι οι πολίτες ιδιαίτερα ε, ακούν με προσοχή και ευαισθησία το μήνυμά σας. Όλα τα μηνύματα, αλλά κυρίως των Γερμανών αδελφών τους η Ένωση βλέπουμε ότι αλλάζει, το Ισλαμικό κράτος βλέπουμε ότι αλλάζει δράση, τρόπο δράσης και δραστηριοτήτων και αφορά αυτό όλα τα κράτη της Ευρώπης και κυρίως επειδή οι τρομοκράτες αναζητούν νέους τρόπους δημοσιοποίησης των δρασίων τους. Μέσα στη δημοκρατική λοιπόν, στο δημοκρατικό γίγνεστη πιστεύετε ότι η διπλωματία της Ευρώπης θα κατευθυνθεί προς νέους προσανατολισμούς ή διαφορετικές στάσεις έναντι ορισμένων κρατών των οποίων θα χρειαστούμε τη βοήθεια για να καταπολεμήσουμε τρομοκρατική απειλή. Επίσης έγινε επίκληση του άρθρου 47 της συνθήκης, 122 για το οποίο έγινε λογότερα λόγος, περί αλληλεγγύης. Δεν είναι όμως και η στιγμή αυτή τώρα η καταλληλότερη για να ξεκινήσει το εγχείρημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας που βρίσκεται στη φασιμότητα εδώ και τόσα χρόνια. Πρόεδρε, πρέπει να πω ότι όπως οι περισσότεροι Ευρωπαίοι έτσι και εγώ αισθάνομαι ότι οδύνει για τις επιθέσεις αυτές εις βάρος των της Γαλλίας. Πρέπει να γίνουν περισσότερα για να προσθεθούν τα σύνορα, για να ενισχυθεί η συνεργασία και βέβαια το, στο διπλωματικό μέτωπο πρέπει πολλά ακόμα να γίνουν. Με ενθαρρύνει το γεγονό ότι κάνατε λόγο για υποστήριξη των δυνάμεων των Πεσμέρκα που καταπολεμούν το Ισλαμικό κράτο. Ε, οι συζητήσει για τη Συρία γίναν και στην Βιέννη πρόσφατα. Μία διάσταση όμω που δεν πρέπει να λησμονούμε είναι ο μουσουλμανικό πληθυσμό τη Ευρώπη. Τα τελευταία πέντε χρόνια μόνο 2% των τρομοκρατικών επιθέσεων στην Ευρώπη οφείλονται σε δράση ε, τρομοκρατικών υποθέσεων, οργανώσεων υποκινούμενων από ιδεολογική ε, βάση και αυτό αφορά η αδίποτε ιδεολογική βάση. Χρειάζεται λοιπόν να λαμβάνονται υπόψη οι θέσεις της αριστεράς και της δεξιάς ανεξαρτήτως πολιτικής ε, προτιμήσεως κατά τρόπον ώστε να αντιληφθεί και ο μουσουλμανικός πληθυσμός στην Ευρώπη ότι τους υποστηρίζουμε και μετά αυτές τις τρομοκρατικές επιθέσεις, οι οποίες τους βγαίνουν τόσες ανησυχίες για ρατσιστικές επιθέσεις και διακριτική μεταχείριση. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ. Παρακαλώ να σέβεστε το χρόνο σας, ο κύριος Νάτ. Πρόεδρε, Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πώς είναι δυνατόν να λέμε ότι αυτή τη στιγμή είμαστε κατά του Ισλαμικού κράτους αφού κάθε στρατιωτικός υπεύθυνο ξέρει ότι το πρώτο που πρέπει να χτυπηθεί είτε είναι η επιμελητία. Αλλά υπάρχουν επτά σημεία επαφή στα οποία διαχειρίζονται το οποιοδήποτε πολεμικό υλικό υπάρχει εκεί στο ε, Κουρδιστάν. Υπάρχουν αυτά τα 7 σημεία, αυτές οι 7 γέφυρες. Ε, αν δεν καταπολεμήσουμε αυτά τα σημεία τι θα γίνει. Επίσης, για το ίσις, 1400 χιλιόμετρα χρειάζεται να έχει το ίσις έδαφος. Μόνο αν ε, βομβαρδίσουμε τα φορτηγά τα οποία μεταφέρουν ε, βενζίνη ε, μπορούμε να χτυπήσουμε πολύ το Ισλαμικό κράτος. Επίσης βλέπουμε να φτάνουν συνεχώς προμήθειες και εφόδια, επίσωτρα, γοκιτόκις, χιλιάδες από το Κατάρ τα έχουν ε, αγοράσει και ε, ε, περνούν μέσω της Κίνας. Τίποτα δεν κάνουμε για όλα αυτά. Πώς λοιπόν θα καταπολεμήσουμε το Ισλαμικό κράτος αν λέει η στρατιωτική στρατηγική ότι χρειάζονται 5,5 χρόνια. Μα είναι αστείο έτσι όπως ακούγεται. παρακαλώ. Εγώ θα αναφερθώ σε δύο ζητήματα που ακροφυγώς έχουν θυγεί και που νομίζω ότι μένουν στη σιωπή. Το ένα είναι η αντίφαση που υπάρχει υποστήριξη προ του πεσμερκά την ίδια ώρα που ξέρουμε ότι η Τουρκία του πολεμά. Και εμεί υποστηρίζουμε όμω από την άλλη μεριά την Τουρκία. Υπάρχει μια αντίφαση που πρέπει να λυθεί. Ο ρόλο του Ισραήλ. Επίση υπάρχει μια μεγάλη σιωπή στο γεγονό ότι αυτά τα δύο κράτη θέλουν να έχουν τη Συρία ένα κράτο δορυφόρο. Και τα αναφέρω διότι είναι δύο ζητήματα που δεν συζητιούνται. Δεν θα αναφέρω τα υπόλοιπα που έχουν λεχθεί. Το δεύτερο, το έχει πει και ο προηγούμενος συνάδελφος, η μεγάλη οικονομική δύναμη του ΝΤΑΕΣ, του Ισλαμικού κράτους, είναι τα πετρέλαια. Δεν χτυπήθηκε καμία φορά ούτε ένα διηληστήριο. Υπάρχει μια απάντηση για αυτό το πράγμα και η τελευταία μου ερώτηση, επειδή ο κύριος Στάιν Μάγερ πάει αύριο στην Κύπρο, θα ήθελα να ξέρω, επειδή υπάρχουν δηλώσεις στην Κύπρο ότι πάει με μια σκέψη υποστήριξης της λύσης, αν έχει κάτι συγκεκριμένο να μας πει. Ευχαριστώ. Thank you. Mr. Thank you. Ευχαριστώ. Λέω ο ε, Κύριε Πρόεδρε, κύριε Υπουργέ, ως επικεφαλής της αντιπροσωπείας για την Ουκρανία, να σας ευχαριστήσω για τα όσα κάνετε στο φόρουμ της Νορμανδίας. Όμως, δεν πρέπει να αποσυνδέουμε βεβαίως τις προσωρινά κατεχόμενες περιοχές του Ντομπάς και την παράνομα προσαρτημένη Κρυμαία σημαντικό αυτό το θέμα. Και δεύτερον, ως συνέχεια των δραστηριοτήτων της ε, Νορμανδίας ε, μπορείτε να σκεφτείτε κάποιες δραστηριότητες επανένταξης των κατεχόμενων περιοχών την πιθανή ανάγκη η διεθνη κοινότητα να ορίσει μια γνωστή προσωπικότητα με στόχο ακριβώς ε, την επανένωση των κατεχόμενων περιοχών. Πρέπει να το σκεφτούμε νομίζω. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κύριε Υπουργέ, για τη Συρία. Μπορείτε να μας δώσετε την αποψή σας για το πώς αξιολογείτε τον ρόλο της ε, Τουρκίας ε, στις σχετικές συνομιλίες που και η ίδια αντιμετώπισε κάποιες επιθέσεις από το Ισλαμικό κράτος και βλέπουμε ε, να επιτίθεται σε κουρδικούς στόχους. Τι προσδοκίες έχετε από την Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας. Εμείς στο Κοινοβούλιο δεν ενθουσιαζόμαστε πάρα πολύ για τη σύνδεση που υπήρξε μεταξύ ε, των συνομιλιών για το μεταναστευτικό με την ένταξη. Συγκεκριμένα αποτελέσματα τι περιμένετε, έχετε ε, μιλήσει με την Τουρκία για ασφαλείς και νόμιμες διόδους ε, για πρόσφυγες. Επίσης η κυρία Μέρκελ είπε πως ε, η συνεργασία θα αυξήσει σε όλους τους τομείς, όχι μόνο στο θέμα των προσφύγων. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ποια είναι η θέση των, της κυβέρνησής σας, ποιοι θα είναι αυτοί οι τομείς της στενότερης συνεργασίας. Βάγγελ και Φλέκενστάιν. Κύριε Βάγγελ Φλέκενστάιν, και τα λοιπά, και ελπί. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ που ήρθατε σε αυτή την συνάντηση. Δυτικά Βαλκάνια. Πολύ σημαντικός επικοδομητικός ο ρόλος της Γερμανίας ε, και για την ανάπτυξη. Αρχή να φέρουμε τη διαδικασία του Βερολίνου, μια πολύ καλή αφετηρία. Πώς βλέπετε το μέλλον ε, της περιοχής αυτής των Δυτικών Βαλκανίων. Βλέπουμε πρόοδο, ενίοτε όμως ε, ανακύπτουν συνεχώς ε, πολιτικές κρίσεις, μια μετά την άλλη σε αυτή την περιοχή. Τι πρέπει να κάνουμε και πού πρέπει να εστιάσουμε για να αποφύγουμε αυτές τις κρίσεις. Ό,τι αφορά τη Σερβία, η μεγαλύτερη πρόκληση της χώρας, ποια είναι για να συνεχίσει με άνοιγμα κεφαλαίων ε, στις διαπραγματεύσεις τις ενταξιακές. Επίσης, σε ό,τι αφορά το μέλλον των διαπραγματεύσεων μεταξύ Κωσυφοπεδίου και Σερβίας, μετανάστευση, είναι θετικό το γεγονός ότι συμμετείχαν στην όλη διαδικασία οι χώρες της περιοχής. Πιστεύετε ότι επαρκεί η πολιτική και χρηματοδοτική στήριξη που τους δίνεται. Ευχαριστώ. Με αλφαγιώτα το δίνετε. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών, ευχαριστώ πολύ για την ομιλία σας και για όσο είπατε για τη φυρία. Από εδώ είναι. Αναφέρατε μόνο στο περιθώριο της ομιλίας σας στην ΤΑΕΣ, ένα από τα εμπόλεμα μέρη. Πώς θα προχωρήσετε από εδώ και μπρος, δεν υπάρχει ο κίνδυνος οι μαχητές του σε περίπτωση ανακοχής να βρουν ελεύθερο πεδίο, ούτως πίν, για να προωθήσουν την κατάκτηση των γύρω περιοχών. Ο κύριος Στόκερ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα πρώτα απ' όλα να εκφράσω την αλληλεγγύη μου από τη θέση αυτή προς τους συναδέλφους Αλιομαρή και Ντόνζο. Έχουμε κι εμείς κήρυξη πένθος στην Ουγγαρία λόγω των επιθέσεων αυτών. Θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω πώς γίνεται να αποφύγουμε την διείσδυση τρομοκρατών στις ροές των μεταναστών. Δεν θα ήταν καλό να ενισχυθεί και η προστασία των συνόρων Σέγγεν με τη Βουλγαρία και τη Ρουμανία, ενώ έχουν αποκλειστεί. Uh, thank you, Chairman. Well, I too uh, wish to uh, share my... Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και εγώ να εκφράσω την αλληλεγγύη μου με τον γαλλικό λαό. Η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω κύριε Υπουργέ, υπό ποιε συνθήκε θα μπορούσε η Γερμανία να στηρίξει και να συμμετάσχει σε μια αποστολή του ΝΑΤΟ κατά του Ισλαμικού κράτους. Ευχαριστώ. κύριε Υπουργέ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να παραμείνω λίγο σε κάποια πλαίσια να απαντήσω πρώτα στο θέμα της Συρίας. Το πρώτο ερώτημα αφορούσε πραγματί το χρονοδιάγραμμα που συμφωνήσαμε το Σάββατο που μας πέρασε, το οποίο οπωσδήποτε είναι πάρα πολύ απαιτητικό. να θυμηθούμε τα του καλοκαιριού που λέγαμε ότι εντός 6 μηνών θέλαμε μια μεταβατική κυβέρνηση και μετά κατάπαυση του πυρός και σε 18 μήνες εκλογές στις οποίες θα μπορούσαν να ψηφίσουν όχι μόνο όσοι βρίσκονται στη Συρία αλλά και οι Σύριοι υπήκοοι της Διασποράς που βρίσκονται και στις ε, χώρες που εκπροσωπούνται εδώ πέρα. Βλέπουμε πως είναι πάρα πολύ φιλόδοξο και απαιτητικό το χρονοδιάγραμμα, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Καθώς για πρώτη φορά όλοι οι εμπλεκόμενοι βρίσκονται γύρω από το ίδιο τραπέζι. Αλλά βεβαίως το θέμα τελικά δεν είναι μόνο το χρονοδιάγραμμα, αλλά και πόσο γρήγορα θα προχωρήσουμε στην ουσία. Και εδώ πέρα πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποιες ε, παρεξηγήσεις που υπάρχουν για το τι εννοούμε όταν μιλάμε για κατάπαυση του πυρός. Ο κύριος Φρόιντ ρώτησε τι γίνεται, πώς εκμεταλλευτεί μια κατάπαυση του πυρός ε, το Ισλαμικό κράτος. Όχι, κοιτάξτε, το έγγραφο της Γέννης εννοεί βεβαίως κατάπαυση των εχθροπραξιών μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολιτευόμενων ομάδων ενόπλων και όπως είπα λοιπόν στις εισαγωγικές μου παρατηρήσεις θα φροντίσουμε να μην μπορέσουν ε, να συγκρουστούν ε, μονάδες ε, του, του στρατού της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης εναντίον ο ενός του άλλου, αλλά να μπορούν να χτυπήσουν τη, το Ισλαμικό κράτος και την ε, Αλνούσρα. Και βεβαίως ε, πρόκειται για μια διαμάχη που έχουμε με την, το Ισλαμικό κράτος και την Αλνούσρα και όχι της ε, δύση ε, με τη Ρωσία ή με κάποιον άλλον. Και βεβαίως βλέπουμε πως ε, και στον αραβικό κόσμο θέλουν να περιορίσουν τον ορισμό των τρομοκρατικών ομάδων στο Ισλαμικό κράτος και την Αλνούσρα, αλλά υπάρχουν άλλοι που λένε πως πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτούς οι οποίοι συνεργάζονται στενά με το Ισλαμικό κράτος. Τελικά το θέμα αυτό, όταν οδηγηθούμε σε αυτή την κατάπαυση του πυρός, θα κριθεί από το ποιος ε, θα συνυπογράψει και θα τηρήσει αυτή την κατάπαυση του πυρός ή όχι. Αυτοί που δεν θα συμφωνήσουν σε αυτήν θα συνεχίσουν να μάχονται στο πλευρό του Ισλαμικού κράτους και οι άλλοι θα ακολουθήσουν μια άλλη πορεία για να θα βοηθήσουν σε αυτή την κατάπαυση του πυρός που περιέγραψα. Τι σημαίνει αυτό για την ε, ευρωπαϊκή αλληλεγγύη. Εγώ συμφωνώ με αυτούς που λένε πως ε, δεν επιτρέπεται να περιοριστούμε μόνο σε δύο λογάκια για την τραγωδία του Παρισιού, αλλά ε, θεωρώ πως όλοι είμαστε σε μια παρόμοια κατάσταση. Η τραγωδία των Παρισιών είναι πραγματικά τρομακτική, αλλά κάποιοι υπενθυμίσατε πράγματι πως υπήρξε και η Μαδρίτη και το Λονδίνο. Γι' αυτό, αυτό το οποίο έχει ήδη ξεκινήσει με βάση τις συνεννοήσεις των Υπουργών Εσωτερικών, οι οποίοι επικοινωνούν και θα συναντηθούν εδώ πέρα την Παρασκευή, είναι ακριβώς η συνεργασία των αστυνομικών αρχών, των μυστικών υπηρεσιών, κάτι το οποίο πλέον είναι κατεπήγον, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν τουλάχιστον οι κίνδυνοι για να αποφύγουμε ανάλογα τέτοια χτυπήματα κάπου αλλού στην Ευρώπη. Αυτό είναι έκφραση της ευρωπαϊκής ε, αλληλεγγύης ε, που εξέφρασαν πάρα πολύ εδώ μέσα. Τώρα, Πώς σχετίζεται αυτό με μια πιθανή στρατιωτική εμπλοκή. Αν όλοι και η Γαλλία ήμασταν πεπισμένοι πως ε, πρέπει τώρα να αναλάβει δράση το ΝΑΤΟ κατά του Ισλαμικού κράτους και της ε, Αλνούστρα, τότε θα ήταν τελείως διαφορετική η κατάσταση. Αλλά θεωρώ πως ούτε η Γαλλία, Ούτε οι άλλες χώρες του ΝΑΤΟ, ούτε ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ θεωρούν πως ε, αυτή είναι μια αποστολή του ΝΑΤΟ και ότι μπορεί το ΝΑΤΟ εδώ να βοηθήσει. Και θα πρέπει να κινητοποιήσουμε τις αραβικές χώρες ε, της Μέσης Ανατολής να εμπλακούν περισσότερο, αλλά όπως σας είπα, όσο καλές και ευχάριστες και ανακούγονται οι προσφορές στρατιωτικών δυνάμεων και μας επενούν τα μήνυε, δεν βοηθούν πάρα πολύ. Η πορεία την οποία πρέπει να ακολουθήσουμε για να μειωθεί το δράμα αυτής της ε, σύγκρουσης και να καταλήξουμε σε μια πολιτική λύση, είναι κάτι που δεν θα το γλιτώσουμε. Οπότε δεν είναι θέμα αριθμού μαχητικών αεροπλάνων ε, ή τεθωρακισμένων, ούτως ή άλλως υπάρχουν πολλά όπλα στην περιοχή, θα πρέπει να επιδοθούμε σε μια προσπάθεια όπως αυτή που περιέγραψα στην εισαγωγή μου. Και να πω και στους Βρετανούς συναδέλφους, στον Βρετανό συνάδελφο, αν η αλληλεγγύη μας μετριέται με το να κάνουμε το ίδιο με αυτό το οποίο έκανε η Μεγάλη Βρετανία. Δεν βοηθάει. Ο καθένας έχει την δική του συνεισφορά. Αν περιοριστούμε όλοι σε αεροπορικές επιθέσεις, για το οποίο προσφέρονται διάφορα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, αν περιοριστούμε όλοι σε αυτό, τότε ισχύει αυτό το οποίο επίσης είπε κάποιος ε, συνάδελφός σας, θα ισοπεδώσουμε την έρημο, αλλά δεν θα σημειωθεί καμία πρόοδος κατά του Ισλαμικού κράτους. Οπότε η απάντηση πρέπει να ανταποκρίνεται στην περιπλοκότητα της κατάστασης. Και η περιπλοκότητα είναι το ότι αυτή τη στιγμή στην Συρία έχουμε ένα πολυμέτωπο πόλεμο. Γίνεται ένας πολυμέτωπος πόλεμος από τον οποίο υποφελείται το Ισλαμικό κράτος. Πρέπει λοιπόν να μειώσουμε τον αριθμό των μετόπων ε, για να πολεμήσουμε πραγματικά το Ισλαμικό κράτος και την Αλληνόσρα. Και όπως σας είπα δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό. Αν θέλουμε να υπάρξει κάποια πρόοδος. Η Γαλλία ε, επίσης ανακοίνωσε πως αν είδα καλά τις ε, ειδήσει από τα πρακτορία θα ακολουθήσει και τον δρόμο του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ και θα ζητήσει εκεί ένα κοινό ψήφισμα με στόχο η αλληλεγγύη αυτή να εκφραστεί και από την κοινότητα των κρατών. Να απομακρυνθούμε τώρα λίγο από το θέμα της Συρίας. Να πάμε στην Τουρκία και τη μετανάστευση. Κάποιος έθεσε το ερώτημα το εάν η Γερμανία είναι διατεθειμένη να επανεξετάσει την πολιτική της και να συνεργαστεί με κάποιες δύσκολες χώρες. Εγώ ήμουν ένας από τους πρώτους που πήγαν στην Τουρκία όταν ε, έγινε σαφής η διάσταση του ζητήματος ε, του προσφυγικού και είπα στον Ερντογάν προσωπικά πως είστε η χώρα κλειδί και πρέπει να βρεθούν τρόποι συνεργασίας έτσι ώστε η ροή τουλάχιστον να είναι προβλέψιμη για τις ευρωπαϊκές χώρες ε, και για εμάς στη Γερμανία άραγε. Ξέρετε πως ο διάλογος για το θέμα αυτό με την Τουρκία συνεχίζεται. Το εάν θα καταλήξει σε ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό για εμάς είναι δύσκολο να το πω αυτή τη στιγμή. Οι προσδοκίες των δύο πλευρών είναι γνωστές. Γνωρίζουμε επίσης πως η Τουρκία πέρα από την οικονομική στήριξη έχει και άλλες προσδοκίες να ξεκινήσουν κεφάλαια των διαπραγματεύσεων και το θέμα της απαλλαγή αποθεωρήσεις. Για εμάς από την άλλη πολλά εξαρτώνται από το εάν η Τουρκία μπορεί να προστατεύσει τα δυτικά σύνορα στην Μεσόγειο για να μπορούμε να γνωρίζουμε πόσοι άνθρωποι έρχονται στην Ευρώπη και βεβαίως αυτό σημαίνει πως ε, και η Τουρκία θα πρέπει να βοηθήσει τους ανθρώπους στο εσωτερικό της για να μείνουν ε, εκεί. Το ερώτημα το οποίο ετέθη για το Αφγανιστάν στο Αφγανιστάν δεν θα βάλουμε κάτι πινακίδες μόνο Προσπαθούμε απλά να καταπολεμήσουμε την προπαγάνδα των διακινητών. Αυτό ισχύει και για το Αφγανιστάν και για πολλές χώρες της Μαύρης Αφρικής που λέει αυτή η προπαγάνδα πως όποιος πάει στη Γερμανία του δίνουν δουλειά, επιδόματα και τζάμπα σπίτι. Να πούμε λοιπόν κάτι για την... να αντιπαλέψουμε αυτή την προπαγάνδα Οπότε ε, γίνεται στα ηλεκτρονικά μέσα, στα ψηφιακά μέσα, στα κοινωνικά δίκτυα και προσπαθούμε να ξεκαθαρίσουμε τις λάθος εντυπώσεις που δημιουργούν οι οργανώσεις των διακινητών. Το εάν τώρα μπορούμε να ξαναστείλουμε κόσμο στο Αφγανιστάν. Αναφέρατε τον Αφγανό Υπουργό Μετανάστευσης, τον Μπάλκι, ο οποίος ε, πράγματι δήλωσε δημοσίως πως όποιος Αφγανός πολίτης έφυγε στο εξωτερικό δεν τον ξαναδεχόμαστε πίσω. Αμέσως ε, εγώ μετά από κάνα δύο μέρες ήρθα σε επαφή με τον Αφγανό πρόεδρο και τον ρώτησα αν ξέρει πραγματικά τις διεθνείς υποκρεώσει της χώρας του. Και το επιβεβαίωσε. Οπότε δεν υπάρχει καμία αλλαγή της ε, νομικής κατάστασης. Το θέμα είναι βεβαίως το τι γίνεται στην πράξη. Όταν θα έχουμε μεγάλες ομάδες ε, Αφγανών ε, που ε, δεν ε, θα λάβουν άσυλο από καμία ευρωπαϊκή χώρα, αν τους στείλουμε πίσω, αν θα τους δεχτούν. Και βεβαίως... Υπάρχει και θέμα βεβαίως με την γερμανική νομοθεσία που λέει πως ε, θα πρέπει πράγματι να βρεθούν περιοχές στις οποίες δεν θα υφίσταται κρατική δίωξη και συνθήκες ε, εμφυλίου πολέμου. Μετά, για το θέμα της Ουκρανίας. και των κυρώσεων. Συχνά με ρωτάνε οι δημοσιογράφοι. Συμφωνείτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την παράταση των κυρώσεων. και μου προξενεί, μου κάνει εντύπωση γιατί εγώ αλλιώ βλέπω την αποστολή μου. Η αποστολή μου είναι να φροντίσω στους υπουργού εξωτερικών να μην υπάρχει ανάγκη για κυρώσει. Οπότε το να επιβεβαιώσω ότι θα συνεχίσουν να είναι αναγκαίες οι κυρώσεις δεν είναι αυταξία. Αν πρέπει λοιπόν να αποφασίσουμε τέτοιες ε, κυρώσεις, αυτό αντικατοπτρίζει μια θλιβερή αλήθεια ότι ε, δεν κάνουμε τίποτα ουσιαστικό. Γι' αυτό να υπενθυμίσω ποια είναι η αποστολή μας στην εξωτερική πολιτική. Είναι να διασφαλίσουμε πως θα συνεχιστεί η διαδικασία του Μίνσκ ε, και γι' αυτό ακριβώς ε, παλεύουμε, σας διαβεβαιώ. Και μετά τα μικρά βήματα προόδου που είχαμε πρόσφατα θεωρώ πως ε, ότι είμαστε σε καλό δρόμο. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε τα επόμενα βήματα εφαρμογής. Και βεβαίως και δεν είναι τίποτα το καινούριο αυτό το οποίο σας λέω, το έχουν συμφωνήσει οι αρχηγοί κρατών το μέλλον των κυρώσεων θα εξαρτηθεί από την εφαρμογή των συμφωνιών του Μίνσκ. Και εάν δεν υπάρχει κάποιος τρόπος για τις Ουκρανικές αρχές ε, να αποκαταστήσουν ε, τον έλεγχο των συνόρων, προφανώς δεν ε, θα έχει εφαρμοστεί πλήρως το πρωτόκολλο του Μίνσκ. Θα ξεκινήσει λοιπόν τώρα η συζήτηση μεταξύ των Υπουργών Εξωτερικών για το πώς θα μπορέσουμε να λάβουμε κάποιες αποφάσεις τον Δεκέμβριο έτσι ώστε το μέλλον των κυρώσεων να εξαρτάται από την εξέλιξη της διαδικασίας του Μίνσκ. Και νομίζω πως το αργότερο τον Φεβρουάριο θα δούμε το εάν οι εκλογές έγιναν με βάση των συμφωνιών των Παρισίων και του Βερολίνου όπως έχει συμφωνηθεί. Εάν είχαν εάν γίνουν οι εκλογές έχουμε κάνει ένα παραπάνω. Έχουμε εκλογές, ε, μια νέα νομοποίηση και βεβαίως μετά θα τεθεί ενισχύ ο νόμος ε, του ειδικού καθεστώτος αλλά ξέρω τι τεράστιο βήμα είναι αυτό γιατί μετά παραμένει ανοιχτό το ζήτημα του πώς ε, θα ανακτήσει τον έλεγχο των ανατολικών συνόρων της η Ουκρανία. Επομένως, αφήστε να γίνει αυτό η συζήτηση σε επίπεδο Υπουργών των Εξωτερικών και να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο μέσα από τη διαδικασία του Μίνσκ και να μην συζητούμε μόνο για κυρώσεις. Να δω λίγο στο κατάλογο. Δυτικά Βαλκάνια έχουν διαδραματίσει ρόλο. Συμφωνώ κύριε Κούκαν. Η διαδικασία του Βερολίνου μας ανέφερε στον ορθό δρόμο και νομίζω και η διαδικασία της προσέγγισης με την Ευρώπη έχει ενισχυθεί. Κατά τη ε, διάρκεια της διαδικασίας του Βερολίνου βέβαια σημειώσαμε και που βρίσκονται τα κύρια προσκόμματα. Ήταν η Γερμανο-Βρετανική πρωτοβουλία η οποία τώρα έχει εξαπλωθεί σε μια ευρωπαϊκή και που προσπάθησε να δώσει, να ξαναξυπνήσει μια δυναμική στη μια Ερσεγοβίνη. Προχώρησε καλά για ένα διάστημα, τώρα παραμένει η απειλή του δημοψηφίσματος με αυτή ζούμε στη Ρεπούμπλικα Σερψκά και ελπίζουμε ότι θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Οι τωρινές εξελίξεις στη Μακεδονία που έχετε βέβαια φαντάζομαι όλοι ε, παρακολουθήσει μας δείχνουν ότι δεν υπάρχει τόση προσέγγιση των Δυτικών Βαλκανίων μεταξύ τους και προς την Ευρώπη. Αντιθέτως, γίνονται όλο και μεγαλύτερες αντιθέσεις μεταξύ τους. Κύριε Κουκάν, ε, για το αν υπάρχει επαρκής οικονομική υποστήριξη. Τους τελευταίους μήνες ε, έχουμε λάβει διαφορετικές και δικρόμενες πληροφορίες. Υπήρξε κάποια εποχή όπου οι πληροφορίες μιλούσαν και από τη Σερβία και ρητά σε συνεντεύξεις τύπου κτλ. Ε, δήλωναν ότι δεν ζητούν λεφτά από την Ευρώπη. Τώρα βλέπουμε να αλλάζει αυτό. Εκ μέρους της Γερμανίας μπορώ να πω ότι ήμασταν το μόνο ε, κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης που συνέχισε να προσφέρει οικονομική υποστήριξη στην Σερβία. Σε ένα βαθμό τουλάχιστον και ξέρετε ότι έχουμε βοηθήσει σημαντικά τη χώρα αυτή. Για την Κύπρο, τελευταίο. Ναι, και τεύτερο ερώτημα. Αύριο όντω θα επισκεφθώ την Κύπρο. Είναι καιρό που δεν έχω πάει. Εάν υπάρχουν κάποια θετικά και ενθαρρυντικά μηνύματα, νομίζω αφορούν αυτή την μακροχρόνια σύγκρουση στην Κύπρο. φαίνεται να υπάρχει επικοδομητικός διάλογος μεταξύ του βόρειου και του νότιου τμήματος της Κύπρου, λέει ο και ελπίζουμε ότι θα οδηγήσει σε μία λύση. Εκείνοι οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν τις αρχές του βορρά και τον νότο φαίνονται πως την έχουν αξιοποιήσει τη δυνατότητα αυτή επιρροής θετικά. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ λέει ο Πρόεδρος. Ευχαριστούμε για τη δυνατότητα να γίνει αυτή η συζήτηση. Μια-δύο παρατηρήσεις αν μου επιτρέπετε. Γιατί πιστεύω ότι πρέπει να παταχθεί το ΙΚΙΛ, το Ισλαμικό κράτος. Είδαμε και την αντεπίθεση των Πεσμέρκα και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει πως υπάρχει δυνατότητα να επιτύχουμε νίκες. Πρέπει να τους απομονώσουμε και να προσφέρουμε την υποστήριξη εκεί που χρειάζεται και βέβαια να διακόψουμε τις ροές των χρημάτων και τις χρηματοδότηση από το πετρέλαιο. Δεύτερον, υπάρχουν πράγματα που δεν πρέπει να αναμειγνύονται ελαφρά την καρδία. Η Ευρώπη βρίσκεται ενώπιον δύο σημαντικών προκλήσεων, την ε, αντιμετώπιση της τρομοκρατίας αφενός, την ε, προσφυγική κρίση εφετέρου. Πρέπει να προσέξουμε να μην αναμειγνύονται στο δημόσιο διάλογο τα δύο αυτά θέματα και να μην ε, ε, να μην γίνεται το αμάλγαμα μεταξύ προσφύγων και τρομοκρατίας. Είναι θύματα της τρομοκρατίας οι πρόσφυγες, δεν έχουν συνάφεια με την τρομοκρατία. Ταυτόχρονα πρέπει εμείς οι Ευρωπαίοι να εργαστούμε μαζί και πρέπει να αντιληφθούμε ότι κανένα ε, κράτος εθνικό δεν μπορεί μόνο του να διαχειριστεί, να αντιμετωπίσει τα προβλήματα αυτά, μικρό ή μεγάλο, και στην τρομοκρατία αλλά και στην προσφυγική κρίση δεν μπορεί κανείς μας μόνος του να τα αντιμετωπίσει. Και η πολιτική βέβαια διαχείριση με τη διαδικασία της Βιέννης που δίνει προγράμματα δράσης νομίζω ότι μπορεί να δώσει λύσεις. Δεν είναι η ώρα τώρα να πούμε ότι έχει αποτύχει η Ευρώπη. Είναι η ώρα αντίθετως να αναγνωρίσουμε ότι χρειαζόμαστε την Ευρώπη για να λύσουμε τις κρίσεις αυτές. Και πρέπει αυτό να καθίσετε πάντα σαφές, ώστε να μην αφήνουμε πεδίο στους ε, λαϊκιστές σε αυτούς που προσπαθούν με μαγικά κόλπα να λύσουν τα προβλήματα. Σας εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία αύριο στην Κύπρο και ελπίζω και εγώ να αναγνωριστεί και να εξασφαλιστεί αυτή η δυνατότητα προσφέρουν οι μοναδικές τα τελευταίες, τελευταίες δεκαετίες ευκαιρίες για διάλογο στην Κύπρο. Ευχαριστώ πολύ. Dear colleagues, could uh, Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Θα συνεχίσουμε με το επόμενο σημείο τη διάταξης, το υπαριθμό 6. Ήτη, την ανταλλαγή απόψεων με τον κύριο Άντριαν Κάντου, πρόεδρο της Μολδαβικής Βουλής, σε σχέση με την πολιτική κατάσταση στη Μολδαβία. Είχαμε μάλλον γίνεται αυτή η συζήτηση σε συνεργασία με την αντιπροσωπεία στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Σύνδεση τη Ευρωπαϊκή Ένωση Μολδαβία. Να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Μολδαβικής Βουλής. Ήταν μια δύσκολη χρονιά για τη Μολδαβία. Η πολιτική κατάσταση στη χώρα ήταν εύθραυστη και στις 29 Οκτωβρίου η κυβέρνηση του Πρωθυπουργού διαλύθηκε διότι δεν πήρε την πρόταση ε, αξιοπιστίας, έγινε πρόταση μορφής στη Βουλή. Μια νέα κυβέρνηση θα πρέπει να σχηματιστεί, δεν έχει γίνει ακόμη αυτό. Θα είναι η τρίτη μέσα στην ίδια χρονιά. Επίσης η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει παράσχει φέτος ε, και πολιτική και οικονομική υποστήριξη γιατί υπάρχει πολιτική κρίση διαρκής που έχει αυξήσει την ε, ε, έλλειψη εμπιστοσύνης των πολιτών στο ότι θα μπορέσει η χώρα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που είναι η καταπολέμηση της διαφθοράς και η μεταρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και της οικονομίας. Αντιλαμβανόμαστε ότι και το τραπεζικό σκάνδαλο που είναι γνωστό ε, είδε τα φώτα της δημοσιότητας πριν από ένα χρόνο αλλά δεν έχει ακόμη ερευνηθεί. Υπάρχουν πολιτικές δυσκολίες ε, που αποτελούν τροχοπέδι ε, για τις διαπραγματεύσεις Είχαμε την προηγούμενη εβδομάδα μια δημοσκόπηση της κοινή γνώμης που δείχνει την κρίση και τη δυσαρέσκεια της κοινή γνώμης με την κυβέρνηση. Φαίνεται λοιπόν ξεκάθαρα ότι ο μολδαβικός λαός αναζητεί και επιδιώκει μια κυβέρνηση, ένα συνασπισμό φιλοευρωπαϊκό ε, και νέες εκλογές. Ανησυχούν οι πολίτες για τη διαφθορά και θέλουν να γίνουν πράξη οι υποσχεθήσει, οι σα μεταρρυθμίσει. Θα δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο του Κοινοβουλίου τη Μολδαβία τον κύριο Κάντου, για να μα ενημερώσει για ένα δεκάλεπτο περίπου σε σχέση με τα σημαντικότερα αισθήματα της επικαιρότητα και τα μέτρα για την αντιμετώπιση των κρίσιμων ζητημάτων που ανέφερα εγώ. Και θα ήθελα επίση να μα πείτε κύριε Κάντου πώ βλέπετε τι εξελίξει στη Μολδαβία δεδομένου ότι είστε ένα από τους σημαντικούς εταίρους ε, στην πολιτική γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κύριε Κάντο, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πλένκοβιτς. Καταρχάς θα ήθελα να πω ότι με τιμά η πρόσκληση. Είναι προνόμιο να βρίσκομαι απόψε εδώ για να σας δώσω τις τελευταίες πληροφορίες για το τι συμβαίνει στη Μολδαβία και βέβαια να έχουμε και μια ανταλλαγή απόψεων και σκέψεων. Η Μολδαβία ήταν μια ιστορία επιτυχίας του προγράμματος γειτονίας. Είχαμε αυτή την ταμπέλα. Δυστυχώς όμως άρχισαν να αντιμετωπίζει διαστατικά προβλήματα και η θετική τάση αυτή χάθηκε σιγά σιγά. Να πω λοιπόν καταρχάς ότι σήμερα δύο λέξεις είναι σημαντικές για να μπορεί κάποιος να κατανοήσει την κατάσταση στη Μολδαβία. Η πρώτη λέξη είναι απογοήτευση. Πράγματι είναι μια μεγάλη απογοήτευση για την πολιτική, υπάρχει μάλλον πολιτική απογοήτευση απέναντι στην πολιτική τάξη εν γέννη και ε, τα κυβερνητικά κόμματα, όλες ιδιαίτερος, λόγω των καθυστερήσεων στις μεταρρυθμίσεις, ε, τις απαιτούμενες ε, θεσμικές μεταρρυθμίσεις, ιδίως για το δικαστικό σύστημα, το τραπεζικό σύστημα και άλλα. Χάσαμε την αξιοπιστία μας, χάσαμε την εμπιστοσύνη των Μολδαβών πολιτών, όπως χάνουμε και την εμπιστοσύνη και αξιοπιστία των εταίρων μας, μεταξύ αυτών και των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Πολλές όμως ήταν και οι θετικές εξελίξεις, τα επιτεύγματα της Μολδαβίας, η οποία επέγραψε και άρχισε την υλοποίηση της Συμφωνίας Σύνδεσης ε, εδώ και ένα χρόνο και έχουμε καλά αποτελέσματα και στο εμπορικό σκέλος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα είναι ο πρώτος εμπορικός εταίρος της Μολδαβίας. Με τη δική σας βοήθεια ε, καταφέραμε και με επιτυχία από τη ρωσική αγορά να περάσουμε στις ευρωπαϊκές αγορές και ιδίως σε μια χρονική περίοδο όπου η Ρωσία επέβαλε εμπάρκο ε, στα προϊόντα από τη Μολδαβία. Επίσης έγινε πολύ σημαντική δουλειά για την υλοποίηση πολλών συγχωνεύσεων και την, συγγνώμη, για την υλοποίηση πολλών μέτρων και για την απελευθέρωση τη των διαφατήρων. Αυτά είναι θετικά. Όμως δεν διαχειριστήκαμε σωστά το τραπεζικό ζήτημα, το οποίο γνωρίζετε. Είχαμε μια υπόθεση διαφθοράς, ε, απάτης και μετά καθυστέρησαν σημαντικές διαφορετικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι το δεύτερο πρόβλημα. Και έχασε την αξιοπιστία της τρέχουσα πολιτική τάξη. Τώρα, δίπλα στην οικονομική την χρηματοπιστωτική κρίση έχουμε και την πολιτική κρίση. Βρισκόμαστε σε συνομιλίες και επαφές για, την, ε, για το σχηματισμό ε, της νέας κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας όσο το δυνατόν πιο σύντομα, ώστε να δοθεί στην ε, κυβέρνηση η αρμοδιότητα και να μπορέσει να ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις ε, για τα επόμενα τρία χρόνια με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο. Μεταξύ των προτεραιοτήτων είναι ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε και να διαχειριστούμε με το σωστό τρόπο. Μεταξύ αυτών είναι τραπεζικός τομέας, Θέλουμε να περάσει νομοθεσία και να εφαρμοστεί ένα σύστημα που θα ε, προσφέρει διαφάνεια σε σχέση με τους μετόχους, ε, την εταιρική διακυβέρνηση και άλλα σχετικά ζητήματα, ανεξαρτησία της Κεντρικής Τράπεζας είναι ένα από αυτά. Το δεύτερο ζήτημα είναι η μεταρρύθμιση ε, του δικαστικού συστήματος στο κοινοβουλευτικό θεματολόγιο. Έχουμε ένα νέο νομοσχέδιο σε σχέση με την πολιτική, με την εισαγγελία σε συνεργασία με την Επιτροπή της Βενετίας και εμπειρογνώμης από την Ευρωπαϊκή Ένωση προχωρούμε το έργο αυτό. Έχουμε λοιπόν και ένα πρόγραμμα αξιολόγηση από ομοτήμου, από ομοτήμου από την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα ελέγξουν ε, του φορεί ε, πολέμηση τη διαφθορά. Έχουμε βέβαια και καλή νομοθεσία, λίγου ε, θεσμού, λίγα θεσμικά όργανα. Κάτι όμω δεν λειτουργεί σωστά, κάτι δεν πηγαίνει καλά. Επίση η ενέργεια είναι προτεραιότητα. Η Μολδαβία εξαρτάται από μία πηγή ενέργειας, ε, ουσιαστικά ρωσική προέλευση, φυσικό πέτρελο και φυσικό αέριο από την Πενιστερία. Θα πρέπει λοιπόν να ε, πιέσουμε τα πράγματα για να υπάρξει μεγαλύτερη διασύνδεση, καλύτερη διασύνδεση της ε, Μολδαβίας με το ευρωπαϊκό ε, σύστημα μέσω της Ρουμανίας. Θέλουμε αγωγούς ε, πετρελαίου και φυσικού αερίου και με αντίστροφη ροή μεταξύ Ρουμανίας και Μολδαβίας, αλλά θέλουμε να βελτιώσουμε και το επιχειρηματικό περιβάλλον, που προτεραιότητα βέβαια είναι να έχουμε και το δικαστικό σύστημα μεταρρυθμίσει και να έχουμε βελτιώσει τον αγώνα μας κατά της διαφθοράς. Σήμερα όμως δεν συζητούμε για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τις σχέσεις που έχουμε σήμερα. Γιατί το μπαλάκι είναι στο δικό μας ε, στρατόπεδο, στη δική μας ε, πλευρά του γηπέδου και πρέπει εμείς πλέον να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. και η προτεραιότητα για την κυβέρνηση η οποία θα σχηματιστεί για την κοινοβουλευτική πλειοψηφία παραμένει και η δέσμευση που έχουμε να λάβει παραμένει η οποία είναι καταρχάς να υλοποιήσουμε την ECFTA, ε, τη Συμφωνία Σύνδεσης. Αυτή είναι η βίβλος μας, αυτός είναι ο γνώμονας που μας καθοδηγεί. Κάθε σελίδα, κάθε κεφάλαιο να εφαρμόσουμε την Συμφωνία Σύνδεσης. Διότι πρόκειται για ε, την εμπιστοσύνη που μπορεί να ανακτηθεί μόνο με συγκεκριμένες δράσεις και ενέργειες και μεταρρυθμίσεις. Ο χρόνος φρέχει και από τα ωραία λόγια και τα μηνύματα πρέπει να περάσουμε στα έργα, στις πράξεις. Και ακριβώς αυτό επιδιώκει η πολιτική τάξη και πρέπει να κάνει στη Μολδαβία, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν θα αποκατασταθεί εμπιστοσύνη της κοινή γνώμης και επομένως ε, η χώρα θα μπει σε μια μακροχρόνια πολιτική κρίση ίσως ε, έλθουν πρόορες εκλογές, ε, αλλά αυτό θα σημάνει το άνοιγμα του κουτιού της Πανδώρας. Κανείς δεν θα ξέρει τι πρόκειται να επακολουθήσει και η επιρροή άλλων χωρών, ιδίως της Ρωσικής Ομοσπονδίας, μπορεί ε, πραγματικά να γίνει αισθητή. Σας ευχαριστώ θερμά που με ακούσατε και τώρα είμαι στη διάθεσή σας να απαντήσω στα ερωτήματά σας. Είναι προνόμιο που βρίσκομαι εδώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε κύριε Υπουργέ για να μπορέσει ο πρόεδρος ε, του Κοινοβουλίου να απαντήσει. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να ζητήσω από την κεφαλής αντιπροσωπείας ε, τον κύριο Κριστέα και τον κύριο Αστοβίτς ε, να μιλήσουν για δύο λεπτά και οι υπόλοιποι συνάδελφοι από ένα λεπτό για να είμαστε εντός του χρόνου και καλωσορίζω και τον επικεφαλής αντιπροσωπείας της Ένωσης ε, στη Μολδαβία, τον κύριο Ταπιόλα που είναι επίσης εδώ. Και ευχαριστώ για τις προσπάθειες που καταβάλλετε στο Κισνόβιον. Κύριε Κριστέα, έχετε το λόγο για δύο λεπτά. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, καλώς ήρθατε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η αντιπροσωπεία μας ανησυχεί ιδιαίτερα από την κατάσταση που υπάρχει στην Μολδαβία και θα ήθελα να πω ξεκάθαρα πως λόγω της ανευθυνότητας των πολιτικών ηγετών που ιδιωτικοποίησαν τα θεσμικά όργανα του κράτους εμείς ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση καταλήξαμε να στηρίζουμε μια δημοκρατία της ε, Μολδαβίας χωρίς ε, μεταρρυθμίσεις. Αυτό είναι λάθος. Θα πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία των μεταρρυθμίσεων στο εσωτερικό της ε, χώρας ε, και βεβαίως ε, στο Κισινάου είχατε μια σειρά ευκαιριών που πλέον δεν υπάρχουν. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει κάνει πολλά όμως για τη Μολδαβία και εξακολουθεί να κάνει. Λαμβάνεται την, τα περισσότερα δάνεια κατά κεφαλήν σύμφωνα με την Συμφωνία Σύνδεσης και πριν από ένα χρόνο και τρεις ημέρες κυρώθηκε και σχετική συμφωνία από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ανησυχώ λοιπόν ιδιαίτερα. Για τα όσα συνέβησαν πριν από δύο ημέρες όταν το PDM καταψήφισε τον κυβερνητικό συνασυσμό στον οποίο ανήκε. Καταψήφισαν την κυβέρνησή τους. Ε, ήταν μια πολιτική ε, χειρονομία λανθασμένη κατά την άποψή μου όσον αφορά την ε, πολιτική του Κισινάου η δικιά μου η εμπειρία είναι πως δεν είναι αφελής και δεν κάνω λάθος υπολογισμούς γι' αυτό ανησυχώ ακριβώ για τη Μολδαβία να πω τώρα κάποια πράγματα για τον κύριο Βορώνιν ο οποίος παρακολουθούσε την εφαρμογή της ε, Συμφωνίας ε, Σύνδεσης είπε πως ε, είμαστε πραγματικά ακατανίκητοι στην διαδικασία αυτή. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Κριστέα. Σας ο εισηγητής. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Επιτρέψτε μου κύριε Πρόεδρε τη ε, Βουλής ναι. τη μολδαβία να σα καλωσορίσω και εγώ ναι. στι Βρυξέλλε. Καλό είναι να έρχεται κανεί στι Βρυξέλλε και πολλέ φορέ καλή αργά παρά ποτέ. Αλλά το γεγονό ότι παραμένουμε στρατευμένοι υπέρ μια ευρωπαϊκής Μολδαβία πρέπει να είναι για εσά βεβαιότητα. Θέλουμε μια ευρωπαϊκή πορεία για την ε, Μολδαβία Ελπίζουμε μετά από κάποιες καθυστερήσεις και σύγχυση η Μολδαβία να μπορέσει να ξαναβρει το δρόμο της και να ολοκληρώσει τη συμφωνία σύνδεσης με όλο το θεματολόγιο που βλέπετε. Αντιλαμβανόμεθα βεβαίω τι σημαίνουν οι μεταρρυθμίσεις, το να ξεκινήσει κανείς μεταρρυθμίσεις ή ακόμα και να χτίσει ένα κράτος. Παίρνει χρόνο, χρειάζεται πολλή βούληση, ακόμη και νέες συμμαχίες πολλές φορές. Και συμφωνώ ότι σήμερα πρέπει να μιλούμε ειλικρινά και απερίφραστα. Άλλη λύση δεν υπάρχει. Κύριε Πρόεδρε της Βουλής Μολδαβίας, ξέρετε πως και εγώ ότι στην πολιτική το 99% της δουλειάς είναι η εμπιστοσύνη. Όλα τα άλλα είναι τεχνική. Πρωτόκολλα, καφέδες κτλ. Είπατε κι εσείς όμως ότι η απώλεια αξιοπιστίας και υποστήριξης είναι το κύριο χαρακτηριστικό της πολιτικής ζωής στη Μολδαβία σήμερα. Θα γνωρίζετε ασφαλώς ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν χρειάζεται άλλη μια ε, ε, περιφερειακή κρίση. Δεν θέλουμε να δούμε τη Μολδαβία να προχωρεί προς την κατεύθυνση αυτή. Δυστυχώς όμως στο στάδιο που βρισκόμαστε μόνο με ερωτήσεις μπορούμε να απαντήσουμε ή με συστάσεις, απαντήσεις συγκεκριμένες δεν μπορούμε να δώσουμε. Ερωτώ λοιπόν τι πρέπει να γίνει για να περιοριστεί στην πολιτική της χώρας σας η επίδραση των ολιγαρχών. Είναι πολύ μικρή η χώρα σας. Δεν είναι δυνατόν να την κυβερνούν ένας, δύο ή τρεις το πολύ ολιγάρχες. Δεύτερον, βλέπετε να υπάρχει κάποια πιθανότητα ε, βράχει πρόθεσμα να ξεκινήσει μια νέα ευρωπαϊκή ε, κυβέρνηση συνασπισμού, φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση συνασπισμού, ώστε να ξαναμπεί στον ορθοδρόμο η Μολδαβία. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κριστιαν Μπρέντα ε, από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε της Βουλής της Μολδαβίας. Σας καλωσορίζω σήμερα εδώ και πιστεύω ότι όπως είπατε και εσείς η δημοκρατία της Μολδαβίας έχει κάνει το αντίθετο από το επίτευγμα. Δηλαδή έχει μέσα ένα χρόνο υπονομεύσει την πρόοδο που είχε μέχρι τώρα επιτύχει. Το αντίθετο από αυτό που θα έπρεπε να επιδιώκεται και θα επαναλάβω την ερώτηση του κυρίου Κριστέα. Έγινε μια έκκληση για το Βορονίν. Εκλήθητε να συμμετάσχετε σε μια νέα κυβέρνηση. Και όλα αυτά μέσα σε πολλές εντάσεις. Συμμαχία λοιπόν, συνασπισμός κυβερνητικός, φιλοευρωπαϊκός. Ένα. Δεύτερον, ο ρόλος των ολιγαρχών και κυρίως του κυρίου Πλαχότνικ που είναι ε, ε, το αφεντικό του πολιτικού σας κόμματος ουσιαστικά. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε ότι υπάρχει δυνατότητα ε, να κρατήσετε φιλοευρωπαϊκό δρόμο με τους ολιγάρχες ή θα πρέπει να τους βγάλετε από τη μέση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Δεμέρξ Μάρκερ είναι εδώ. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. πέσατε το των τύπων των ήλων είπατε πως ε, χάθηκε η εμπιστοσύνη στους ε, πολιτικούς. Και βεβαίω εμεί στηρίζουμε την Μολδαβία στον αγώνα κατά της διαφθοράς ε, και υπέρ των δημοκρατικών αξιών. Και βλέπουμε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση πραγματικά δεν πρέπει να απομακρυνθεί από τις καρδιές των ανθρώπων στη Μολδαβία. Λοιπόν, η Ευρώπη παρουσιάζεται θετικά στα ΜΜΕ. Και ποιος είναι ο ρόλος των Ρώσων και της ρωσικής προπαγάνδας. Ένα άλλο θέμα για τις μειονότητες που θα μπορούσαν να μπλοκάρουν οι γκαγκαούζοι στο νότο παραδείγματο χάρη δεν είναι ικανοποιημένοι με το ρόλο που παίζουν στη Μολαβία και ζητάνε στήριξη από τη Ρωσία. Πώς θα δώσουμε περισσότερο λόγο στη μειονότητα αυτή για να έχουμε μια πιο διευρυμένη κυβέρνηση. Και τέλος, μπορέσατε να παρακάμψετε το ρωσικό εμπάργο κατά της χώρας σας και να αντισταθμίσετε με τη Συμφωνία Σύνδεσης ε, τα προβλήματα που αυτό σας δημιούργησε. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο στοχευμένο εμπόριο με τα κλασικά σας προϊόντα, το κρασί και τα κρέατα κτλ. Thank you very much, Mark. Now I give... Ευχαριστώ, Μάρκ. Η κυρία Γκάμπριελ Τσίμερ έχει τώρα το λόγο. Ja, vielen Dank. Ε, ευχαριστώ. Είπαμε πως σκοπεύετε να μεταρρυθμίσετε το σύστημα της δικαιοσύνης για να καταπολεμήσετε την διαφθόρα. Σωστό αυτό. Το θέμα είναι ποιος θα το κάνει. Γιατί δημιουργείται η εντύπωση πως η πολιτική τάξη η ίδια είναι διεφθαρμένη και έχει εμπλακεί σε τραπεζικά σκάνδαλα. Θα ήθελα λοιπόν να μάθω σε ποιο βαθμό συμπεριλαμβάνεται εδώ πέρα και τον πόλεμο κατά της φτώχειας. Ξέρουμε πως η Μολδαβία είναι μία από τις φτωχότερες ευρωπαϊκές χώρες και νομίζω πως για να ξανακερδίσει η πολιτική τάξη στην εμπιστοσύνη αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να γίνει. Και θα ήθελα μετά να γνωρίζω εάν τμήμα της μεταρρύθμισης ε, της δικαιοσύνης είναι το τι γίνεται με τους πολιτικούς κρατούμενους εξ όσων γνωρίζω και μπορείτε να μου πείτε αν ισχύει ή όχι είναι δυνατόν να κρατήσει η προφυλάκηση μέχρι και 6 χρόνια. Έξι χρόνια στη φυλακή χωρίς να πάει κανείς ε, στο δικαστήριο. Να πω επίσης πως τις ε, διαδηλώσεις ε, της 6ης Σεπτεμβρίου συνελήφθησαν πάρα πολλοί άνθρωποι μεταξύ των οποίων ο πρόεδρος ε, του Κόκκινου Μπλοκ, ο Γρηγόρη Πετρένκο που είναι μέλος επίσης της αντιπροσωπείας ε, του Μολδαβικού Κοινοβουλίου με το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και υπήρξε αίτημα του Συμβουλίου της Ευρώπης να αφαιθούν ελεύθεροι συλληφθέντες και να τους αντιμετωπίζεται δίκαια τι σκοπεύετε να κάνετε εδώ. Ευχαριστώ, Κάρβερ; Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ ειλικρινής. Όταν έγιναν πέρυσι εκλογές στη Μολδαβία, 21% και 25 έδρες κέρδισε το Ευρωσκεπτικιστικό κόμμα και έγινε το μεγαλύτερο κοινοβουλευτικό κόμμα. και τώρα προσπαθούν να σχηματίσουν κυβέρνηση από κοινού ε, τα κόμματα του φιλοευρωπαϊκού συνασπισμού. Τον Απρίλιο μόνο 32% των Μολδαβών είναι υπέρ της σύνδεσης. Αυτό λέει μια σφιγμομέτρηση. Το 2007 το ποσοστό ήταν συντριπτικά υπέρ. Μεγάλη πτώση Θέλω να μας πείτε, η Μολδαβική κυβέρνηση ε, αναγνωρίζει ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο τμήμα πλέον του μολδαβικού πληθυσμού που δεν θέλει. Μας είπε ο κύριος Γιούνκερ επίσης ότι δεν θα υπάρχει διεύρυνση τα επόμενα πέντε χρόνια. Υπάρχουν διασφαλίσεις πολιτικές ή θεσμικές για την ε, δίκαιη ε, διαβούλευση με τους Μολδαβούς πολίτες αν η Μολδαβία αποφασίσει να ξεκινήσει ε, πενταξιακές συζητήσεις. Ευχαριστώ. Σόλτς, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ και για τα σχόλιά σας. Πριν από τρεις εβδομάδες ε, περίπου είχαμε την τρίτη συνεδρίαση της Εμπορικής Επιτροπής ε, όπου ετέθη εκεί το θέμα της FTA, της συμφωνίας που βρισκόμαστε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο επίσης συζητεί ένα νέο νομοθέτημα για τις ασφαλιστικές δικλείδες ε, επί του παρόντος. Εσείς αναφερθήκατε σε ορισμένα προβλήματα ε, πολιτικά και δικαστικά ζητήματα που ανακύπτουν. Θα ήθελα να μας δώσετε λίγο περισσότερες λεπτομέρειες και να είστε λίγο πιο συγκεκριμένος. Πώς θέλετε να στηρίξετε τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων υπάρχουν κάποιες πτυχές της DCFTA που δεν έχουν εφαρμοστεί ακόμη συζητάμε τα επόμενα βήματα. Δεν θα πρέπει όμως να μας πείτε λίγο περισσότερα για να γνωρίζουμε πού βαδίζουμε, πού βρίσκεται η συνεργασία και στο εμπορικό σκέλος, γιατί αυτό επηρεάζει και την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της χώρας. Όχι μόνο ε, τους φορολογούμενους ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, επηρεάζει τους πολίτες της δικής σας χώρας κυρίως. Πρέπει να υπάρξει ε, μια ομαλή ε, εξέλιξη στη χώρα σας και μια ισορροπημένη κοινωνικο-οικονομική εξέλιξη και ανάπτυξη. Ο κύριος Πλένκοβιτς, ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον πρόεδρο της Μολδαβικής Βουλής, τον κύριο Κάντου, ο οποίος στα επόμενα 5-6 λεπτά θα προσπαθήσει να απαντήσει σε όλες τις ερωτήσεις. Ευχαριστώ, θα προσπαθήσω να είμαστε το δυνατόν πιο σύντομο. Θέλω να σας ευχαριστήσω για όλες ε, τις ερωτήσεις και να μου επιτρέψετε να δώσω έμφαση σε ένα πολύ σημαντικό σημείο χαιρετίζουμε και αναγνωρίζουμε την πολύ σημαντική ε, υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για όλα όσα έχουν γίνει στη Μολδαβία ό,τι αφορά την απευθέωση καθώς θεωρήσεων, ε, την συμφωνία σύνδεσης, τα κτλ. Παραλαμβάνω ότι τώρα εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να δράσουμε για να αποκαταστήσουμε την εμπιστοσύνη και για να τρέξουμε τις μεταρρυθμίσεις. Τώρα, σε ό,τι αφορά την υλοποίηση της, της FTA, Υπάρχει πρόοδο, το 15% της συμφωνίας της FTA ήδη έχει εφαρμοστεί, υλοποιείται. Όμως, εν γέννη συμφωνία σύνδεσης της FTA δεν είναι πια ένα ζήτημα εξωτερικής πολιτικής, αλλά είναι πια ένα ζήτημα εσωτερικής εθνικής πολιτικής. Θα εστιάσουμε τις προσπάθειές μας λοιπόν σε, στη συγκρότηση μιας ειδικής ομάδας αντίστοιχο με ένα Υπουργείο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων. Θα είναι ένας φορέας ε, που θα συσπηρώνει τι προσπάθειε όλων των φορέων ε, της ε, συμφωνίας σύνδεσης και της, της συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου. Στη σύντομη ιστορία μας για πρώτη φορά πλέον έχουμε ένα θεματολόγιο με προτεραιότητα την ε, υλοποίηση της συμφωνίας των άρα ξέρουμε ακριβώς τι πρέπει να γίνει κάθε φορά. Έχουμε χρονοδιαγράμματα και προθεσμίες, ε, είναι οι αρμόδιοι και συναρμόδιοι ε, σε δράση και όλοι θα είναι υπόλογοι και για την υλοποίηση αλλά και για την μη υλοποίηση ενδεχομένως, Στις καθυστερήσεις δηλαδή που ίσως προκύψουν. Σίγουρα πρέπει να γίνει δουλειά και νομοθετική δουλειά αλλά και εφαρμογή των νόμων που θα περάσουν και δεν θα είναι εύκολο αυτό. Μπορώ να σας πω ότι στο Κοινοβούλιο συζητούμε ε, το νέο νομοσχέδιο για την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο, για την ενέργεια, ούτω ώστε να έχουμε το δεύτερο και το τρίτο ενεργειακό πακέτο. Αυτά μόνο σε εθνικό επίπεδο μπορούμε να τα πετύχουμε. Σε ό,τι αφορά τις φυσικομετρήσεις ε, και την ε, αξιοπιστία κτλ. Και την άποψη των πολιτών για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Επειδή δεν πετύχαμε στις μεταρρυθμίσεις και επειδή υπήρξε και η ρωσική προπαγάνδα, πράγματι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχασε, πώς να το πω, υποστηρικτές μεταξύ του μολδαβικού πληθυσμού, αλλά αυτό δεν οφείλεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά γι' αυτό ευθυνόμαστε εμείς και τα δικά μας σφάλματα. Και η ρωσική προπαγάνδα ευθύνεται. Διότι κάποιος ε, μίλησε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πόσο ισχυρός είναι ο αντίκτυπος των μίντια και των ρωσικών σταθμών. Είναι μεγάλος ο αντίκτυπος, μεγάλη επιρροή. Πάνω από τα μισά τηλεοπτικά κανάλια είναι ρωσικά. και όταν έχουμε και το ευρύτερο περιφερειακό πλαίσιο που δεν έχει να κάνει μόνο με τη Μολδαβία, καταλαβαίνετε. Πρέπει να σας πω ότι ο κόσμος βλέπει πολύ τηλεόραση. Η τηλεόραση είναι η βασική πηγή ενημέρωσης για το πολύ κόσμο και επηρεάζει πολύ. Αν με ρωτήσετε πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε αυτή την πρόκληση, μόνο με δημοκρατικό τρόπο είναι η απάντηση. Δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε τους ρωσικούς σταθμούς, τα ρωσικά κανάλια. Δεν είναι αυτό ελευθεροτυπία, δεν είναι αυτό ελευθερία λόγου. Υπάρχουν άλλα μέτρα όμως. Και το πρώτο θα ήταν να προωθήσουμε και να βοηθήσουμε την ανάπτυξη των τοπικών προϊόντων. Με ειδικά προγράμματα, με το ΞΟ για την Ευρωπαϊκή Ένωση, πόσο σημαντική είναι και λεγόμενες κοινωνικές διαφημίσεις. Η κοινωνία εν γέννη και η πολιτική τάξη και το κοινοβούλιο συζητούν πλέον νομοσχέδια, παραδείγματος χάρη. Πρώτα απ' όλα, να έχουμε διαφάνεια και στην ιδιοκτησία των μίντια. Δεύτερον, πρόθεση ανάπτυξη τοπικών προϊόντων για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις λόγω της ρωσικής προπαγάνδας. Ρωσικό εμπάργκο. Η παραγωγή οι γεωργοί, οι κτηνοτρόφοι της Μολδαβίας πλήττονται ε, τα μάλα από το ρωσικό εμπάργο και θα τους πάρει χρόνο μέχρι να μπορέσουν να καταληφθούν τις νέες αγορές. Διότι δεν έχουν την απαιτούμενη γνώση, εμπειρία, ούτε και τα απαιτούμενα κονδύλια. Είναι πολύ δαπανηρό. Πώς θα πάρει κανείς ε, δάνειο όταν ε, το επιτόκιο μπορεί να είναι 20% στη Μολδαβία σε σχέση με τους παραγωγούς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως, Νομίζω ότι εξελίσσεται γρήγορα ο κόσμος και μεταπηδεί από τη ρωσική στην ευρωπαϊκή αγορά. Και εμείς σίγουρα θα στηρίξουμε όσο μπορούμε αυτή τη μετακίνηση. Σε ό,τι αφορά τις μειονότητες και την ένταξη των μειονοτήτων. Όπως γνωρίζετε, στο νότιο τμήμα της χώρας ε, έχουμε αυτονομία για τους καγκαούσους. As well as to have a communication on... Προσπαθούμε να προωθήσουμε την επικοινωνία. Και στο επίπεδο της κυβέρνησης ε, και του Κοινοβουλίου. Εγώ έχω υποβάλει μια πρόταση, η οποία ελπίζω σε 15 μέρες να εγκριθεί για μια σύσταση μιας ομάδας εργασίας μεταξύ του Ομοσπονδιακού Κοινοβουλίου και του τοπικού κοινοβουλίου της Γκαγκαουζίας της αυτόνομης περιοχής για να βρεθεί μια λύση και στα θέματα τα νομοθετικά. Ένα συνάδελφος ρώτησε για το θέμα της ε, κράτησης ε, στο πλαίσιο της δικαιοσύνης. Ε, εγώ από όσο γνωρίζω κρατείται κανείς μόνο 30 μέρες συν να παραταθεί για άλλες τόσες. Έξι χρόνια δεν υπάρχουν αυτά που λέτε. Μετά υπάρχει μια δίκαιη δίκαιη όπως θα γίνει και στην περίπτωση Πετρένκο άλλωστε. Το παρακολουθεί και το Συμβούλιο της Ευρώπης και εμείς παρακολουθούμε το θέμα αυτό. Οπότε προηγείται όπως είπα η δίκαιη δίκη και το κράτος δικαίου. Μετά ετέθη ένα ζήτημα για τους ολιγάρχες και συνολικά για το πώς επηρεάζουν τα θεσμικά όργανα. Δεν έχει σημασία το όνομα κάποιου, αυτό το οποίο έχει σημασία, είναι τα θεσμικά όργανα. Οι, θεσμοί, για να απαντήσω λοιπόν τώρα στα ρουμανικά. Μεγάλη μου λύπη διαπίστωσα πως δεν ήμασταν σε θέση να οικοδομήσουμε αξιόπιστα θεσμικά όργανα τα οποία θα φροντίσουν να υπάρξει μια σταθεροποίηση. Αν δούμε τα δυτικά, λειτουργεί το σύστημα, λειτουργούν οι νόμοι και όσο πιο πολύ πάμε στα ανατολικά της χώρας, ε, τόσο πιο πολύ μπαίνει θα έλεγα ο ανθρώπινος παράγοντας. Υπάρχουν αιτήματα, τηλεφωνήματα κτλ. Πρέπει λοιπόν να δημιουργήσουμε ένα σύστημα στο οποίο θα λειτουργεί ο νόμος και να μην έχει σημασία το εάν κάποιος είναι ολιγάρχης ή όχι. Έτσι θα αλλάξει η πολιτική ατζέντα στη Μολδαβία και τότε δεν θα μιλάμε για τα ονόματα και τα και για το ότι κάποιος έχει περισσότερη επιρροή από άλλους χρειαζόμαστε θεσμικά όργανα τα οποία θα λειτουργούν στο προσεχές μέλλον θα γίνουν αυτές οι μεταρρυθμίσεις ε, τις οποίες ε, περιμέναμε για να δημιουργήσουμε θεσμούς που δεν θα επηρεάζονται από κανέναν ούτε και από τους ολιγάρχες. Και βεβαίως ο κύριος Κριστέα μετά έθεσε το ζήτημα πιθανού συνασπισμού με τους ε, κομμουνιστές. Κοιτάξτε. Εγώ ανήκω σε μια νέα πολιτική γενιά και ειλικρινά σας λέω εγώ φυλάγομαι όταν ακούω κομμουνιστές και το τι σημαίνει αυτό λόγω και του παρελθόντος. Δεν ξέρω αν μπορούμε να συνεργαστούμε με ένα ακόμα όταν δεν τηρεί και τις ε, δεσμέσεις του. Π.χ. αυτά από και την συμφωνία σύνδεσης. Αυτή τη στιγμή λοιπόν μπορούμε να επιτύχουμε κάποια πλειοψηφία χωρίς ε, τις ψήφους των κομμουνιστών, αλλά φοβάμαι πως τον Απριλίο που θα πρέπει να εκλέξουμε πρόοδο θα Εξαρτώμεθα από τους ε, κομμουνιστές και κάποια στιγμή βεβαίως θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με την εμπλοκή του Κομμουνιστικού Κόμματος. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε ποιος θα εκλεγεί πρόεδρος ε, της Δημοκρατίας της Μολδαβίας Μπορεί να είναι κάποιο ο οποίο δεν θα έχει σχέση με την πολιτική, μπορεί να είναι κάποιος πανεπιστημιακό παραδείγματο χάρη. Έτσι θα έχουμε κάνει ένα πρώτο βήμα για να δημιουργηθεί μια κυβερνητική πλειοψηφία. Αλλά βεβαίως θα πρέπει να υπάρξει ένας ε, συμβασμός των πολιτικών κομμάτων στη χώρα για να εκλεγεί πρόοδος στο Μάρτιο τον Απρίλιο. Τον πρόεδρο βεβαίως τον εκλέγει το κοινοβούλιο και έτσι ίσως ε, οδηγηθούμε σε νέα πολιτική κρίση και νέες εκλογές. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε για την ενημέρωση αυτή, για τις δηλώσεις σας, για τις μελλοντικέ μεταρρυθμίσεις Τελειώσαμε λοιπόν με αυτό το σημείο της ημερησίας διάταξης. Θα ψηφίσουμε σε δύο λεπτά. Dear colleagues, I apologize. Αγαπητοί συνάδελφοι, το συγγνώμη για την σύντομη καθυστέρηση, αλλά ξέρετε ότι έτεινε ούτω ή άλλω να πάει για 6,5 ψηφοφορία όλο το απόγευμα. Πριν όμω ξεκινήσουμε τι ψηφοφορίε, ο κύριο Πρέντα ζητάει το λόγο για τεχνικό ζήτημα. Ναι, Πρόεδρε, πολύ σύντομα γιατί είναι πολλέ ψηφοφορίε. Είχαμε ένα πολύ λυπηρό επεισόδιο κατά την ανταλλαγή απόψεων με τον Υπουργό από τη Γεωργία. Εκπρόσωπος της ομάδας του κυρίου Λεπένα χαρακτήρασε τον Υπουργό της Επιτροπής, τον Πρόεδρο της Επιτροπής των Εξωτερικών Υποθέσεων αλήτη βουαγιού. Είναι πολύ λυπηρό αυτό και καλό τους συναδέλφους από τις άλλες πολιτικές ομάδες να συζητήσουμε το θέμα σε μια ειδική συνεδρίαση ώστε να εξετάσουμε τι είδους μέτρα μπορούμε να λάβουμε εναντίον τη ομάδα αυτή, η οποία δεν σέβεται ούτε τη διαδικασία ούτε και το ύφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Βεβαίω λέει ο πρόεδρο, ευχαριστώ πάντα τα σώμεθα υπέρ του σεβασμού μεταξύ συναδέλφων. Αγαπητοί συνάδελφοι, έχουμε μακρά, ε, μακρύ κατάλογο ψηφοφοριών. Ξεκινώ με την πρώτη έκθεση. Σχέδιο εκθέσεως για τις εξαγωγές όπλων, εφαρμογή κοινή ε, θέσεως. 89-44, Μποντήλ Μπορέρου. Θέλει κάτι ο συζητητής. Η συγγετρία, παρακαλώ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τους κοιόδης συζητητές. Ήταν επικοδομητικές οι συζητήσεις. Καταλήξαμε νομίζω συμβαστικά ότι μπορούμε να έχουμε μια ευρεία πλειοψηφία σε έναν κόσμο όλο και πιο ανασφαλή είναι πολύ σημαντικό να ελέγχονται οι ήρωε ε, του εμπορίου των όπλων, ώστε να μην καταλήγουν σε λάθο χέρια, τα οποία μετά θα να χτυπήσουν εμάς εδώ στην Ευρώπη. Υπό το φως των πρόσφατων ε, επιθέσεων στο Παρίσι, τη Βηρητό και άλλες γειτονικέ χώρες, κάθισε αυτή η ανάγκη πιο σαφής ακόμη. Ξεκινήσαμε από διαφορετικές θέσεις και θεωρήσει, και μπορέσαμε εν τέλει να καταλήξουμε σε κάτι στο οποίο μπορούμε όλοι να συμφωνήσουμε. Αναγνωρίζοντα τη νέα κατάσταση τη σχετική με την ασφάλεια που αντιμετωπίζουμε, αλλά και το ρόλο που έχει δραματίσει στο παρελθόν η βιομηχανία των όπλων για τι νέε εξελίξει και την τεχνολογία βέβαια. Ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε ευρύτατη συνένεση για την έκθεση. σα. ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Βαλέρο. Αρχίζει η ψηφοφορία συμβαστική. μόνο ένα παρακαλώ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. 37 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές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 κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 94 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η τροπολογία 99 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 100 υπέρ. Κατά αποχές απερίφθη 101 υπέρ κατά αποχές θα πρέπει να την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά νομίζω παρακαλώ πρόκειται για την 101 Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 107 με προφορική τροπολογία την υπαριθμό 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 112 να επαληθεύσουμε επαληθεύουμε την 108 Είχατε δίκιο. Εγκρίθηκε, λέει ο πρόεδρος. Ω, με συγχωρείτε, όχι. Απερίφη. Ε, άρα είχα δίκιο την πρώτη φορά. Με ξάφνιασε που κατάλαβα πως έχω άδικο. Λοιπόν, πάμε, αφού απερίφθη 108, στην 112 υπέρ. Κατά. Αποχές, απερίφθη. 111 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 110 υπέρ κατά αποχές πρέπει να επαληθεύσω 110 Απερίφθη. 109. Όχι, 113 λέει ο πρόεδρος. Παρακαλώ. Α, όχι. 109, ε, υπέρ. Κατά. Κατά. Αποχές απερίφθη. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές. Πρέπει να επαληθεύσουμε. Πάλι φαίνεται ένα μοιρασμένο ψήφι. Εγκρίνεται. 114 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας επαληθεύσουμε. Εγκρίνεται. 115 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 117 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 118 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε παρακαλώ. Εγκρίνεται. 123 υπέρ. 123 υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 134 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 135 υπέρ. Κατά Αποχές. Απερίφθη. 136 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 137 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απερίφθη. Συμβιβαστική 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 16 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 154 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 155 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 156 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 157 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 158 υπέρ κατά ας επαληθεύσουμε παρακαλώ 158 εγκρίνεται 19, συμβαστική 19, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. «164 με προφορική τροπολογία την υπαριθμόν 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». «Συμβαστική 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται». «168 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 169 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 170 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 171 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 176 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 177 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 178 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 179 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 180 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 181 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται αιτιολογική σκέψη 5, τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές απερίφθη α με 6 υπέρ κατά αποχές απερίφθη Α, νέο 7 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται ΑΒ νέο 10 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται το Β. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται 12 υπέρ με και τροπολογία την υπαριθμών 2 αποχές εγκρίνεται συμβαστική 22 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και λογική σκέψη δέλτα 14 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε Θεωρητική σκέψη D, τροπολογία 14 εγκρίνεται. Η 15 τώρα υπέρ, κατά, αποχές. Να επαληθεύσουμε. Δεν σηκώνεται όλο το χέρι και είναι πιο δύσκολο έτσι το έργο μας. Στη 15 παρακαλώ επαλήθευση. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. D, ε, Μητροπολογία 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, αιτιολογική αναφορά 14 με τη 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 3 στην 20, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Επαληθεύουμε. Σωστά είπαμε. Εγκρίνεται προφορική τροπολογία υπερθμών 1 υπέρ, κατά, αποχές και εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά η ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε. εγκρίνεται. 52 ψήφοι υπέρ, 6 ψήφοι κατά και 6 εποχές. Συγχαρητήρια στην εισηγήτρια. Την ευχαριστούμε. Και περνάμε στην επόμενη έκθεση Τη κυρία. Πρόκειται για μια ε, έκθεση για μη νομοθετικό ψήφισμα σε απόφαση του Συμβουλίου, των Συμπερισμάτων του Συμβουλίου για τη Συμφωνία Πλαίσιο Συνολικής εταιρική Σχέσης και συνεργασίες μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της αφενός και της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας του Βιετνάμ αφετέρου με εισηγήτρια την κυρία Μπάρμπαρα Λόχφιλερ. Θέλετε να γράψετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω τους ε, σκιώδεις εισηγητές. Είχαμε πάρα πολύ επικοδομητική συνεργασία στι περισσότερες συμβαστικές προτάσει, Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ συμβαστική 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 42 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 45 υπέρ κατά αποχές. Μοιάζει σαν να απορρίφθηκε να την επαληθεύσουμε. 45. Εγκρίνεται. Λοιπόν, ψηφίζουμε τις 46 ε, και 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτές Τροπολογία 50 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 51 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ κατά αποχές δεκτή 54 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά εποχές 59 θα έλεγα απορρίπτεται να την επαληθεύσουμε 59 59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 γραμματεία εδώ πέρα μου λέει πως πρέπει να... με τι ψηφίζουμε. Λοιπόν, 58. Με συγχωρείτε. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Την 64 να την επαληθεύσουμε. Ε, εγώ βλέπω καλύτερα από εδώ πάνω. Συνδυαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 69 ε, υπέρ κατά εποχές απορριφθείτε συμβαστική 6 υπέρ κατά εποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβιβαστική 8 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 83 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή Τροπολογία 91 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 92 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 93 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 94 μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτό. Μέρος δεύτερο υπέρ. Σηκώστε το χέρι παρακαλώ για το δεύτερο μέρος της 94. Κατά. Αποχές. Σαν να απορρίφθηκε μου μοιάζει. Απορρίφθηκε. Απορρίφθηκε. Συμβιβαστική 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 97 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 100 υπέρ κατά αποχές δεκτή 101 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 12 χωριστή ψηφοφορία υπέρ του πρώτου μέρους κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές Δεκτό. 105 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 13 υπέρ. Κατά. Με συγχωρείτε πρέπει να ψηφίσουμε την 106 γιατί απορρίφθηκε η 105. 106 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 110 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 111 υπέρ. Κατά. Αποχές απορριφθείται. 113 υπέρ κατά αποχές δεκτή 112 υπέρ κατά αποχές σαν να απορρίφθηκε να επαληθεύσουμε την 112 Κάποιος δεν ψήφισε. Να εγκρίνεται. 114 υπέρ, κατά αποχές δεκτή, 115 υπέρ, κατά αποχές εγώ θα έλεγα απορρίπτεται, αλλά δεν σηκώτα και τα χέρια. Τι θέλετε, να τα επαληθεύσουμε, να τα επαληθεύσουμε. Κουράζεστε, κουράζεστε. Δεν ψηφίζουν όλοι. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 14 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 119 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 120 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 121 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 122 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 123 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 124 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 100, ε, συμβαστική 16 ε, υπέρ κατά αποχές δεκτή, 125 υπέρ κατά αποχές απορρίφθηκε 130 υπέρ κατά αποχές δεκτή 132 υπέρ κατά αποχές δεκτή 133 υπέρ κατά αποχές δεκτή 134 υπέρ κατά αποχές δεκτή νομίζω δεν ξέρω αν ο κύριος Φλέκενστάιν σηκώνει το χέρι, είναι όλοι, αριστερά από εκεί. Ε. Ναι, μπορούμε να την επαληθεύσουμε. 134. Δίκιο είχα λοιπόν. Ε, μα... Μόνο ο κύριος θα σηκώνει τα χέρια από 37 άτομα. Εγκρίνεται λοιπόν. 135 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 100. Όχι. 1. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 2 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτό. 3 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή, 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 11 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 12 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ, κατά αποχές να την επαληθεύσουμε γιατί δεν σηκώνεται το χεράκι. Πέρασε λοιπόν, εγκρίνεται. 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προφορική τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 16 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές δεκτή η ηλεκτρονική ψηφοφορία στο σχέδιο έκθεσης όπως τροποποιήθηκε παρακαλώ ψήφισαν όλοι κάποιος δεν ψήφισε ακόμα εγκρίνεται ευχαριστώ πάρα πολύ συγχαρητήρια στην κυρία Λοχμπίλερ Περνάμε τώρα. Για την ε, συμφωνία πλαίσιο με τη ε, Δημοκρατία του Βιετνάμ κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονικά είπατε πρέπει να το ψηφίσουμε. Ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά για να καταγραφεί και στα πρακτικά. Για το Βιετνάμ το σχέδιο σύστασης. Υπέρ, κατά, λέει ο πρόεδρος. Okay, thank you. Ευχαριστώ, εγκρίνεται. Τώρα έχουμε την έκθεση της κυρίας Καλνιέτη. Για τη πρωτοκόλλου συνεργασίας για την αληθή υπόψη προσχώρηση της Δημοκρατίας Κροατίας στην Ένωση. Δεν ξέρω αν θέλει πει κάτι η Σάντρα, ας ψηφίσουμε ηλεκτρονικά καλύτερα. Πέρας, πέρας. Εγκρίνεται. Να ευχαριστήσουμε τη Σάντρα και να περάσουμε τώρα στο σχέδιο γνωμοδότησης για την κατάσταση στην περιοχή της Μεσογείου και την ανάγκη για μια ολιστική προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση. Εισηγητής ο Δημήτρη Παπαδάκης. Θέλετε να πείτε κάτι. Θέλω να ευχαριστήσω τους και όλους εισηγητές για την καλή συνεργασία. Θα προσπαθήσω να συμπεριλάβω όλα τα σημαντικά στοιχεία. Σας ευχαριστώ. Thank you, Mr. Ευχαριστώ κύριε Παπαδάκη. Συμβαστική 1 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ. Κατά αποχές <clears throat> εγκρίνεται. Τροπολογία 23 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 4 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 56 κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα ψήφι υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπλία 58 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 77 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 81 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 7 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 103 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 104 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται 105 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 8 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 9 υπέρ, κατά,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 εγκρίνεται. Συμβιβαστική, όχι, ναι, συμβιβαστική 11, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 145 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 146 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 148 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβαστική 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 154 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται 157 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 163 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 165 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 166 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 167 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προφορική 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται προφορική 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται ηλεκτρονική τώρα ψηφοφορία του συνόλου της τροποποίησης εκθέσεως Thank you very much, Mr. ευχαριστώ πολύ κύριε Παπαδάκη. Συγχαρητήρια. Και ερχόμαστε στην τελευταία έκθεση για απόψη. Σχέδιο έκθεσης ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, ετήσια έκθεση. ο Κρίστιαν Πρέντα. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Θέλω να ευχαριστήσω τις πολιτικές ομάδες για την συνεργασία τους ιδίως ό,τι αφορά την ιδέα να είναι βανάγνωστη σύντομη η έκθεση. Γι' αυτό και έχουμε 48 συμβιβατικέ προτάσεις. Αυτό το πλαίσιο λυπούμε λοιπόν, που η Επιτροπή Γυναικών ήθελε να συντάξει μια γνωμοδότηση που ήταν πιο μακροσκελή από την ίδια την έκθεση. Αλλά τέλος πάντων θα την περικόψουμε κάπως, θα την ψαλιδίσουμε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Σεγητά. Να συγκεντρωθούμε για να έχουμε τελειώσει με αυτή την ψηφοφορία πριν τι 7.30. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Αποχέ, εγκρίνεται. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 8 υπέρ. Κατά απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 96 υπέρ. Κατά αποχές ελέγχουμε. Εγκρίνεται. Τροπολογία 97. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 98 υπέρ. Α, συγγνώμη, συγγνώμη, συγγνώμη, ταυτόσημες έχει εγκριθεί μαζί με την 97. 99 υπέρ, κατά, αποχές. Δεν σηκώνετε τα χέρια. Οπότε ή θα πιστεύω το κύριο Φλέκενστάιν ή πρέπει να επαναλαμβάνουμε. Λοιπόν, τώρα επαναλαμβάνω το 99. Υπέρ, κατά, αποχές. Να ελέγξουμε. Ναι, γιατί δεν με παρακολουθήσατε. Λοιπόν, ηλεκτρονικός έλεγχος, άρχεται. That's why I couldn't tell. Γι' αυτό. Δεν μπορούσα να καταλάβω. 30 υπέρ, 28 κατά. Εγκρίνεται. 101 υπέρ, κατά. Αποχές. Ελέγχουμε και για αυτήν. Εγκρίνεται. 112 υπέρ, κατά. Συγγνώμη, 102 διορθώνει ο πρόεδρος. 102 υπέρ Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 103 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 104 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 105 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 106 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 107 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 108 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 9 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 111 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 10 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 116 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 119 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 120 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 11 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 125 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 126 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 128 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 12 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 133 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 138 υπέρ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 156 υπέρ, κατά, αποχές, ελέγχουμε την 156, άρχεται η ψηφοφορία. Α, δεν σηκώνετε τα χέρια σας. 157 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 18 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 162 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 163 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 164 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβαστική 19 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 169 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 20 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 198, τρία τμήματα, πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ. 198, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ. Α, καταπίπτει, μάλιστα, συγγνώμη. Δεν το ψηφίζουμε αυτό. Το τρίτο τμήμα το ψηφίζουμε ή όχι. 198 τμήμα τρίτο. ψήφι υπέρ. Κατά. ΠΟΧΕΣ, Απορρίπτεται. Αφού δυσκώνετε τα χέρια σας. Με δυσκολεύετε. Να επαναλάβουμε ηλεκτρονικά την ψηφοφορία επί του τρίτου τμήματος της 198 τροπολογίας. Απορρίπτεται. Άρα καλά τα έλεγα εγώ. 173 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 174 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Συμβιβαστική 21 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 22 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 183. Περ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 184. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε παρακαλώ την 184. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 25 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 199 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβαστική 26 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 208 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβεβαστική 27 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 214 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Να ελέγξουμε. Απορρίπτεται. Τροπολογία 215. Κατά τμήματα. Πρώτο τμήμα. Ψήφι περ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Να ελέγξουν παρακαλώ. Απορρίπτεται. Τροπολογία 222. Υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 223 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 224 υπέρ. Κατά. απόχέ εγκρίνεται. 225 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 226 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 228 υπέρ κατά αποχές να ελέγξω παρακαλώ. Adopted. Εγκρίνεται. 229 υπέρ κατά αποχές παρακαλώ σηκώνετε τα χέρια γιατί θα πρέπει να ελέγχουμε και γιατί καθυστερούμε και ελέγχουμε και σε αυτή την περίπτωση 229 229 Τρεις δεν την έχουν ψηφίσει ακόμη. Δύο, ένας, πέρας. Έγινε δεκτή. 34 υπέρ. 2.30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 2.32 υπέρ. Κατά. Αποχές να ελέγξουμε. 2.32. Rejected. Απεριφθεί 237 υπέρ 2, 3, 7 υπέρ Ζητώ συγγνώμη, πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία του κυρίου Πρέντα, καθώς η προηγούμενη δεν είχε εγκριθεί. 233 λοιπόν, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 237 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 238 προφορική τροπολογία υπερθυμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 239 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 245 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 256 υπέρ κατά αποχές ε, περίφθη, 257 υπέρ κατά αποχές σαν να εγκρίθηκε. Αλλά ας το επαληθεύσουμε. 257. απερίφθη. 258 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη 259 σε τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 30 ε, υπέρ. Σεβαστική 30 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 262 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε. Εγκρίνεται συμβαστική 31 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 266 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 271 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 272 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 273 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 274 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 33 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. ...283 υπέρ, κατά αποχές απεριευθεί, 287 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 34 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 35 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 307 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 36 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 315 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 317 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 322 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 323 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 324 υπέρ κατά αποχές Επολυθεύουμε. Rejected. Απερίφθη 325 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 326 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται 327 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 39 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 336 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 337 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 340 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 341 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 342 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 443 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 445 υπέρ, κατά αποχές επαληθεύουμε. Εγκρίθηκε 346 υπέρ, ηλεκτρονικά παρακαλώ, μάλλον θα έχουμε το ίδιο. Αποτέλεσμα 346 ηλεκτρονικά. Άλλος ένας, μένει να ψηφίσουν, κλείνει ψηφοφορία και απερίφθη. Συμβαστική 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβαστική 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 43 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 363 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 364 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 44 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 370 υπέρ, κατά. 370 παρακαλώ υπέρ. 370 υπέρ κατά αποχές. απέριφθη 371 υπέρ κατά. απέριφθη 372 υπέρ κατά. Συμβαστική 45 υπέρ κατά. Αποχές εγκρίνεται. 377. υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 378 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 379 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 380 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 382 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε 382. Rejected. Compromise. Απερίφθη συμβαστική 46 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 384 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 385 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 389 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 47 συμβαστική υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 400 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 305 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 307 υπέρ κατά αποχές και επαληθεύουμε Απερίφθη με μια ψηφοδιαφορά 408 υπέρ κατά αποχές επαληθεύουμε 408 εγκρίνεται 409 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 410 4, 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 411 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 412 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 413 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 314 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, συμβαστική 48 υπέρ κατά εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. Αιτιολογική α31 τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, αιτιολογική α, α τροπολογία 34 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 34 την είπαμε, 35 33 λέει ο πρόεδρος. Επαληθεύουμε τη 33. Close. In favor. Adopted 34 in favor. Η 34 έγκρινε υπέρ κατά αποχές. Υιοθετείτε φαντάζομαι, αλλά βλέπω ότι δεν ακολουθούν τα χέρια σας. 34 ηλεκτρονικά. Αχα. Πρέπει να κάνουμε διάλειμμα μάλλον. 35 υπέρ. Κατά. Απερίφθη 36 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 37 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 38 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική υπαριθμών 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 48 υπέρ, κατά αποχές απερίφθη, 49 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 50 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, 51 υπέρ, κατά αποχές επαληθεύουμε, 51. Απερίφθη. Μισοψηφία. 52 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 υπέρ. Κατά. Αποχές και επαληθεύουμε. 53. Εγκρίνεται μια ψηφοδιαφορά. 54 υπέρ. 54 υπέρ κατά αποχές. Τους οριστές 54. Άντε, να το ξαναπούμε. 54 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 3 υπέρ ε, εγκρίνεται. 61 υπέρ κατά αποχές συγκρίνεται 62 61 επαληθεύουμε και έγκρινεται 62 υπέρ κατά αποχές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 84 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. Εγκρίνεται λέει ο πρόεδρος. 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Υπαριθμόν 1 στην αιτιολογική αναφορά υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, υπαριθμόν 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 5 υπέρ εγκρίνεται, 6 υπέρ εγκρίνεται, 7 υπέρ εγκρίνεται, 8 υπέρ εγκρίνεται, 9 υπέρ εγκρίνεται, 10 υπέρ εγκρίνεται, 11 υπέρ εγκρίνεται, 12 υπέρ εγκρίνεται, 13 υπέρ εγκρίνεται, 14 υπέρ εγκρίνεται, 15 υπέρ εγκρίνεται, 16-17 υπέρ εγκρίνεται, 18 υπέρ εγκρίνεται, 19 επίσης, 20 υπέρ 20 υπέρ εγκρίνεται, 21 υπέρ εγκρίνεται, 22 υπέρ Ποια. Ποια θέλετε. Μάλιστα. 20 υπέρ. Κατά. Να την επαληθεύσουμε λοιπόν. Επαληθεύουμε ηλεκτρονικά την 20. Εγκρίνεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 22 υπέρ κατά απορρίπτεται 23 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 23 να την επαληθεύσουμε λοιπόν. Εγκρίνονται. 24 ε, υπέρ κατά εγκρίνεται 25 υπέρ κατά εγκρίνεται 26 υπέρ κατά απορριφθετά 27 υπέρ κατά απορριφθετε 28 υπέρ κατά να την επαληθεύσουμε 28 Αχα. Απορρίπτεται. 29 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Γνωμοδότηση της ΔΕΒΕ. 1. Υπέρ. Κατά απορρίπτεται. 3 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 5 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 6 υπέρ, εγκρίνεται. 7 χωριστή ψηφοφορία, μέρος πρώτο υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο, υπέρ, κατά. Αποχές να την επαληθεύσουμε. Μέρος δεύτερο. ΔΕΒΕ 7. Εγκρίνεται με δύο ψήφους διαφορά. ΔΕΒΕ 8. Όχι, όχι. Συγγνώμη, καταπίπτει. συμφωνείτε να τις ψηφίσουμε όλες από τις ΔΕΒΕ 2 μέχρι τη 12. Ηλεκτρονικά όμως. Απορρίπτονται. Γνωμοδότηση της Επιτροπής Γυναικών. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές. Οι σοσιαλιστές δεν ψηφίζουν. Γνωμοδότηση των γυναικών υπέρ. Α, τώρα εγκρίνεται. 29 υπέρ. Εγκρίνεται. 30 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 31 υπέρ. Εγκρίνεται. 33 υπέρ. Δεκτή. 38 υπέρ, δεκτή. 42 υπέρ, δεκτή. 44 υπέρ, δεκτή. 45 υπέρ, δεκτή. 40 καταπίπτει. 50 υπέρ, εγκρίνεται. 51 υπέρ, εγκρίνεται. 53 υπέρ. 53 υπέρ, υπέρ, κατά, α, εγκρίνεται. 54 υπέρ, κατά, εγκρίνεται. 59 σε δύο μέρη, μέρος πρώτο υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Μέρος δεύτερο υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Μέρος τρίτο υπέρ, κατά, εγκρίνεται. Τέταρτο υπέρ, κατά, εγκρίνεται πέμπτο μεσφαίρ εγκρίνεται. Προτείνουμε να ψηφιστεί unblock οι εξή τροπολογίε τη Επιτροπή Γυναικών. Όλες μέχρι το τέλο, ηλεκτρονικά, αν συμφωνείτε, παρακαλώ. Η Ηλεκτρονική ψηφοφορία για το σχέδιο ψηφίσματος όπως τροποποιήθηκε υπέρ. Ηλεκτρονική. Άλλη μία. Κάποιος δεν ψηφίζει. Είναι σημαντική ψηφοφορία. Εγκρίνεται συγχαρητήρια κύριε Πρέντα. No. When do we Wednesday? we meet Wednesday at 11.30. Very much for your patience. Please remember we have an extra... Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Έκτακτη συνεδρίαση Τετάρτη με τον Επιτροπό Χάν και την κυρία Μογκερίνη. 11 η ώρα. Τετάρτη ευχαριστώ.